Ξεκινάμε και πάλι κυρίες και κύριοι. Σόζα Βάγνερ, εισηγητής. Έχετε το λόγο. 45 λεπτά έχουμε στη διάθεσή μας για να ασχοληθούμε το κείμενο αυτό. Ο εισηγητής 5 λεπτά στη διάθεσή του διαθέτει. Ακριβώς. Ναι, όπως το είπε η κυρία Πρόεδρος, ακριβώς αυτό έχουμε σαν θέμα. Ουσιαστικά πρόκειται για μια γνωμοδότηση η οποία θα πρέπει να σταλεί στην Επιτροπή Περιβάλλοντος και θα αφορά την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την τροποποίηση της οδηγίας 2003 ε, ε, του 87 που διέπει το χρονοδιάγραμμα των πληστηριασμών δικαιωμάτων εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου. Στόχος βασικός ε, είναι το πεδίο εφαρμογή ε, και οι άλλες διατάξεις ε, που αφορούν τους πληστηριασμούς. Δεν νομίζω ότι χρειάζεται εδώ ενώπιον των συναδέλφων βουλευτών να επεκταθώ ιδιαίτερα γιατί το τονίζουμε διαρκώς για το πόσο δηλαδή μεγάλη σημασία έχει η εμπορία αυτή των ε, δικαιωμάτων εκπομπών θερμοκηπιακών αερίου. Πόση μεγάλη σημασία έχει για την Ευρωπαϊκή Ένωση αυτή η πολιτική και σε ό,τι αφορά τον έλεγχο και την προστασία κυρίως του περιβάλλοντος αλλά και όσο έχει να κάνει με την ε, μεταμόρφωση της ευρωπαϊκής βιομηχανίας και του ενεργειακού συστήματος προς μια οικονομία χαμηλών εκπομπών ε, διοξιδίου του άνθρακα. Υπάρχουν και άλλα εργαλεία, αλλά αυτό είναι ένα από αυτά. Είναι ένα από τα εργαλεία που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την επίτευξη των στόχων της βιομηχανικής πολιτικής και της περιβαλλοντικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επαναλαμβάνω και επιμένω ότι ε, δεν χρειάζεται να το τονίσω καν γιατί όλοι έχουμε επίγνωση της σημασίας που έχει πρόταση αυτή της Κομισιόν. Αυτό λοιπόν που προτείνει η Κομισιόν είναι απλά και μόνο να αλλάξει το χρονοδιάγραμμα αυτών των ε, πληστηριασμών δικαιωμάτων εκπομπών. Δεν υπάρχει άλλο στόχος. Αυτό είναι ε, και αποσκοπεί η Κομισιόν με την πρότασή της. Και φαίνεται ότι προκύπτουν κάποιες αμφιβολίες. Σε σχέση δηλαδή με το αν αυτή η πρόταση τροποποίηση χρονοδιαγραμματος της Κομισιόν συμμορφώνεται και με το όλο καθεστώ ε, τη εμπορία δικαιωμάτων εκπομπών θερμοκηπιακών αερίων, διότι πρόκειται για ένα καθεστώ το οποίο έχει δημιουργηθεί γύρω από την ιδέα τη ε, ελεύθερη αγορά. Δηλαδή η αγορά είναι ελεύθερη να δράσει και να καθορίσει και τι τιμέ. Αυτή είναι η βασική ιδέα η οποία εμπνέει και διέπει την ε, εν λόγω αγορά. Πάντως είναι σαφές ότι η λειτουργία της αγοράς αυτής, ε, συνεπία της οικονομικής κρίσης ε, την οποία βιώνουμε, αντιμετωπίζει κάποιες αλλαγές που ανησυχούν ιδιαίτερα, όχι μόνο την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά και όλους τους φορείς που δραστηριοποιούνται στην αγορά αυτή. Οι τιμές έχουν εκτοξευθεί, ε, έχουν πλέον καταλήξει ε, να είναι πιο... Έχει καταλήξει προτιμότερο το να μολύνει κανείς ε, από το να αγοράζει αυτά τα δικαιώματα. Και υπάρχουν και όλες οι πτυχές που σας προανέφερα. Τώρα λοιπόν, στο βαθμό που η αγορά αντιμετωπίζει αυτές τις αλλιώς αυτές τις αλλαγές, έρχεται να παρέμβει ακριβώς εδώ η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Υπάρχει κάποια γενική ένσταση. Ναι, υπάρχει ότι παραδείγματο χάρη, ωραία. Αλλάζει η αγορά, Ας αλλάξει. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα γιατί έτσι γίνονται τα πράγματα, υπάρχουν κάποιοι γενικοί κανόνε, είναι ελεύθερη η ε, τιμολόγηση, ο καθορισμό των τιμών. Δεν είναι μόνο αυτό όμω, υπάρχουν και άλλε επιπτώσει. Δηλαδή, δεν δρούν με αυτόν τον τόσο ξεκάθαρο διαφανή τρόπο, με ελεύθερη προσφορά ζήτηση, όλες οι αγορές, νομίζω ότι είμαστε αρκετά μεγάλοι όλοι για να προβληματιστούμε όταν βλέπουμε μια αγορά να ε, υφίσταται αυτές τις παρεμβάσεις από τη δημόσια εξουσία. Είναι κάτι που το βλέπουμε. Και ιδίω πρέπει να πούμε ότι αυτή η αγορά των, ε, της εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών είναι μια τεχνητή αγορά που τη δημιούργησε η δημόσια εξουσία. Δεν είναι φυσική αγορά, την έχει δημιουργήσει τεχνητά η δημόσια εξουσία και έχει συγκεκριμένους στόχους. Αποσκοπεί σε συγκεκριμένα πράγματα. Επομένως, η βασική ιδεολογική, αν μπορώ να τη χαρακτηρίσω, ένσταση για την αλλαγή αυτών των ε, κανόνων ε, του παιχνιδιού στην αγορά τη συγκεκριμένη, έχει και μια απάντηση ότι δηλαδή περισσότερες αγορές βιώνουν τέτοιου είδους αλλαγέ τη λειτουργία τους Άρα δεν θα πρέπει αυτό να μας φοβίζει. Αν όμως οι γενικοί στόχοι τους οποίους επιδιώκουμε είναι στόχοι που μας βρίσκουν σύμφωνοι και συνάδουν με την περιβαλλοντική πολιτική και την βιομηχανική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επο, επομένως, για να συνοψίσω, βέβαια όλα αυτά θα τα ε, συζητήσουμε και άλλες ε, φορές σε αυτή τη διαδικασία της ανταλλαγής απόψεων. Θέλω να ακούσω τους συναδέλφους μου και τους και ηγητέ βέβαια, αλλά και όλους τους υπόλοιπους συναδέλφους βουλευτέ. Θέλω να ακούσω την άποψή τους για αυτό ε, το θέμα. Και να σας πω από τώρα ότι ο στόχος μου είναι να στηρίξουμε αυτή τη μεταρρύθμιση, την πρόταση δηλαδή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αυτή είναι η δική μου πρόθεση, αλλά φυσικά θέλω να ακούσω τους συναδέλφους. Σας ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Συνάδελφος Τζόρνταν από το ΕΛΚ για τρία λεπτά έχει το λόγο. ναι, Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα ήθελα και εγώ να στηρίξω αυτά τα οποία είπε ο εισηγητής, ότι δηλαδή η Κομισιόν προτείνει έναν ρυθμιστικό μηχανισμό, μα ότι θα είχαμε ένα μηχανισμό αγοράς. Πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί. Υπάρχουν πολλά ζητήματα εδώ κατά την άποψή μου. Πρώτα απ' όλα, λειτουργεί το σύστημα αυτό. Κάποιοι λένε πω δεν λειτουργεί γιατί οι τιμέ είναι πολύ χαμηλέ. Μα οι τιμέ είναι χαμηλέ λόγω τη οικονομική κρίση. Άλλοι λένε πω δουλεύει και πω αυτό είναι ένα φυσιολογικό αποτέλεσμα. Και ε, βοηθάει να επιτύχουν τους στόχους του 2020 κατόπιν. Ε, είναι αυτό ένα κίνητρο για επένδυση σε βιώσιμες τεχνολογίες. Όχι γιατί η τιμή του άνθρακα είναι πολύ χαμηλή και οι πιθανοί επενδυτές δεν έχουν κίνητρο να κάνουν ε, επενδύσεις. Επόμενο ερώτημα μπορούμε να έχουμε την πολυτέλεια να πληρώσουμε κάτι τέτοιο ενώ υπάρχει ακόμα οικονομική κρίση. Και ε, όχι μόνο αυτό, αλλά θα συνεχιστεί η ύφεση. Επόμενη ερώτηση. Ποια είναι η σωστή, θα λέγαμε, η τιμή του άνθρακα. Εάν είναι υψηλότερη κάποια στιγμή στο μέλλον, θα την περιορίσουμε και στο, ως προς το μέγιστο. Επίσης πρέπει να δούμε μια διαφορά μεταξύ εθνικής και ευρωπαϊκής παρέμβασης, γιατί κάποια κράτη-μέλη προσπαθούν να επιβάλλουν τα δικά τους μέτρα. Θέλω να τονίσω και πάλι πως πρόκειται για ένα μηχανισμό της αγοράς, αλλά πρέπει να φροντίσουμε να λειτουργεί σωστά. Πρέπει λοιπόν να κάνουμε κάτι, αλλά η παρέμβασή μας πρέπει να είναι προσωρινό μέτρο. Δεν πρέπει να μειώνει την ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής αγοράς, γιατί έτσι θα χαθούν δουλειές. Επίσης, το ζήτημα δεν είναι τεχνικό αλλά και πολιτικό. Οπότε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει να το παρακολουθεί. Επίσης πρέπει να αρχίσουμε να σκεφτόμαστε τις μακροπρόθεσμες μεταρρυθμίσεις του συστήματος αυτού μετά το 2020 γιατί το σύστημα μπορέας να καλύπτει τους ε, τομείς ενέργειας ε, γιατί στον τομέα της ε, ενεργείας ε, καταλαβαίνετε πως οι επενδύσεις είναι σε βάθος δεκαετιών. Δεν είναι σωστά λοιπόν τα βραχυπρόθεσμα μέτρα. Πρέπει να μιλήσουμε για μεταρρυθμίσεις λοιπόν του συστήματος και μετά το 2020. Ευχαριστώ κυρία Χολ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Το σύστημα αυτό είναι ένας μηχανισμός αγοράς, αλλά δεν υπάρχει πουθενά ένας μηχανισμός καθαρής αγοράς και όπως είπαμε ήδη υπήρχαν κάποια ζητήματα που μείωσαν την τιμή του άνθρακα αρκετά. Είχαμε την οικονομική κρίση που σήμανε μείωση της βιομηχανικής παραγωγής. Είχαμε αναδιάρθρωση σε πολλές ανατολικές χώρες. Είχαμε την μεταφορά υπολείπων αδειών από τη φάση 2 στη φάση 3 και κάποια από αυτά τα πράγματα ήταν καλά από μόνο τους. Αλλά είχαν το αποτέλεσμα να μειωθεί η τιμή. Υιοθετήσαμε μέτρα περισσότερης ενεργειακής αποτελεσματικότητας με τη σχετική οδηγία. Και είχε αναγνωριστεί εκεί πως ε, αυτό θα οδηγούσε την Κομισιόν στο να αξιολογήσει ξανά το ζήτημα των αδειών γιατί θα μπορούσε να επηρεάσει την ε, τιμή του άνθρακα. Και επίσης βεβαίως ε, πουλήθηκαν ε, κάποιες άδειες νωρίτερα για να χρηματοδοτηθεί το πρόγραμμα NER300. Οπότε υπάρχει ένα πλεόνασμα 1,5 δισεκατομμυρίου ή 2 δισεκατομμυρίων αδειών και έχουμε μια τιμή του άνθρακα γύρω στα 10 ευρώ τον Τόνο. Ε, δεν λειτουργεί άρα όπως σκοπεύαμε το σύστημα γιατί στόχο είχε να δώσει κίνητρα για επενδύσεις χαμηλού άνθρακα. Ε, κάποιοι λένε έχει καμιά σημασία αυτό γιατί είμαστε σε σωστή πορεία με τους ε, στόχους μας. Αλλά ακόμα και μία μικρή ανάλυση δείχνει πως ε, παρά, αυτά συμβαίνουν παρά το σύστημα αυτό, παρά την τιμή του άνθρακα και αυτό το οποίο δεν βλέπουμε από τη βιομηχανία είναι ένα μακροπρόθεσμο μήνυμα πως υπάρχει η ανάγκη τέτοιας επένδυσης και είδαμε επενδύσεις σε άνθρακα να αυξάνονται πέρσι γιατί δεν υπάρχει ακριβώ πίεση από το σύστημα αυτό. Η η μηχανία μπορεί να μην έχει δυσκολίες να επιτύχει το στόχο του 2020, αλλά πρέπει να δει παραπέρα το 2030 και το 2050. Και αν είναι χαμηλή η τιμή του άνθρακα, δεν έχουν ένα πλαίσιο για να συμβεί κάτι τέτοιο. Οπότε θεωρώ πως πρέπει να κάνουμε το σύστημα να δουλεύει όπως θέλαμε και να φροντίσουμε η τιμή του άνθρακα να αυξηθεί. Αυτό το οποίο θα έλεγα τέλος είναι πως δεν θεωρώ πως τώρα είναι η ώρα να κάνουμε μεγάλη συζήτηση. Μην το κάνουμε θέμα τώρα, είναι απλό. Απλή η πρόταση της Κομισιόν. Απλά είναι για να υπάρχει νομική βεβαιότητα και το να αλλάξει μόνο το χρονοδιάγραμμα δεν θα επηρεάσει πολύ την τιμή του άνθρακα. Η Κομισιόν θα πρέπει να προτείνει περαιτέρω μέτρα και ελπίζω να το κάνει σύντομα. Η δική μου έκκληση είναι να το τελειώνουμε αυτό εδώ πέρα, να μην, μην, το αρνούμαστε τώρα με τροπολογίες και τελικά συμφωνώ με τον εισηγητή πως πρέπει να στηρίξουμε την Κομισιόν στην πολύ απλή αυτή νομική πρόταση. Ευχαριστούμε. Ζαντό. Merci, Madame la Présidente. Κυρία Πρόεδρε, ευχαριστώ. Κάπως με εκπλήσει αυτό. Αυτή η αγορά των ποσοστώσεων είναι κλασική ιδιωτικού τομέα και όσο γίνεται λιγότερο παρεμβαίνει το κράτος, ε, το δημόσιο, για να μπορέσει να λειτουργεί σωστά. Δεν υπήρχε αυτή η αγορά χωρίς ρύθμιση. Ρύθμιση, αυτή η ρύθμιση δημιούργησε την αγορά. Και όχι την αγορά που χρησιμοποιήσαμε για να ρυθμίσουμε, αλλά αυτή τη ρύθμιση και όλοι μας τι διαπιστώνουμε, ότι δεν λειτουργεί αυτή η αγορά. Ακριβώς ε, αυτές οι ενδείξεις ε, από το δημόσιο που τη δημιούργησε δεν είναι οι σωστές ενδείξεις, τα σωστά σημάδια, σήματα. Ε, εδώ εντάξει έχουμε την κρίση τώρα τα άλλα, αλλά τι μας λέει η κρίση, ότι είναι ο άνθρακας η τιμή του πολύ χαμηλή, δεν είναι της σημερινή αγοράς, αλλά απλά και μόνο για ενόψη μιας μελλοντική ρύθμισης. Και με την κρίση λοιπόν θα έχουμε το 20% της μείωσης των εκπομπών αερίων ε, ε, αερίων θερμοκηπίου. Όχι για τη φιλοδοξία έτσι να ε, λειτουργήσουμε σωστά και όσον αφορά τις ποσοστό, αλλά επειδή με την κρίση θα είμαστε περίπου στο 20% το 2020 της μείωσης των αερίων θερμοκηπίων. Εδώ ε, προχωράμε ακριβώς, είμαστε στη μέση της όλης προσπάθειας και είχαμε ορισμένα συμπεράσματα ε, από ε, από την Τόχα που μας δείχνουν πως έχει τα πράγματα. Και εδώ θέλουμε να δούμε μια καινοτόμα αγορά με τις εκτιμήσεις που έχουν γίνει για το πώς πολλούνται αυτές οι ποσοστώσεις με 30 ευρώ η τιμή του ανθρακ και από εκεί γεννήθηκαν όλες οι εξαιρέσεις. Είμαστε στα 200 δισεκατομμύρια σε 7 χρόνια σε, σε ευρωπαϊκά έσοδα. Τώρα που θέλουμε ε, ίδιους πόρους μέσα χρηματοδότησης, στον αντάλλο για αυτή η μετάβαση ενεργειακή, Ακριβώς θα πρέπει να τα σκεφτούμε αυτά τα πράγματα. Πώς θα είναι αποτελεσματική αυτή η αγορά και για εμά, του πράσινου, του οικολόγου. Θεωρούμε σαφώς ότι η ρύθμιση αυτή της αιτίας θα πρέπει να προχωρήσει ταχύτερα και ότι η αγορά αυτή θα μπορούσε να μας προσφέρει αποτελέσματα, αλλά θα πρέπει ιδιαίτερα να ρυθμίσουμε τις καταστάσεις αυτές. Έχουμε εκατοντάδες εκατομμύρια τόνους υπερβολικού διοξίδου του άνθρακος και γνωρίζουμε όλοι μας ότι δεν είναι αυτό το τμήμα των όσων ε, συζητάμε τώρα, αλλά μετά τι ζητάμε. 1,4 δισεκατομμύρια τόνοι διοξείδου του ε, θα πρέπει να του διαχειριστούμε όπω πρέπει αυτού ε, και μετά από πού περνάει η κατάσταση για να μπορέσει να λειτουργήσει καλύτερα αυτή η αγορά, να δώσουμε τι σωστέ ενδείξει, να περάσουμε σε ένα στόχο 30% τη μείωση τη εκπομπή διοξείδιου του το 2020 και με ένα οδικό χάρτη μέχρι το 2050. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα ήθελα να σα υπενθυμίσω το πλαίσιο των αποφάσεων. Ε, καθώ υπάρχει εδώ πέρα ένα ιστορικό. Το 2008 καταλήξαμε σε ένα πολύ δύσκολο συμβιβασμό στον τομέα της κλιματικής πολιτικής. Ήταν πάρα πολύ δύσκολο για κάποιες χώρες ε, να συμφωνήσουν σε αυτόν τον συμβιβασμό και για κάποιες βιομηχανίες ε, στην Ευρώπη. Και κάποιες από αυτές τις εγκαταστάσεις, τις βιομηχανίες προσαρμόστηκαν στον εαυτό βάρος, ε, κάτι το ήταν πολύ οδυνηρό και κατέληξε στο να μειώσει το επίπεδο επενδύσεων. Και μετά είχαμε επίσης νέα μέτρα και σταθμά και τώρα θέλουμε να το κάνουμε ακόμη πιο αυστηρό γιατί θα αποκλείσουμε 900 ε, εκατομμύρια άδειες και βεβαίως θα υπάρχει μια νέα αλλαγή σε δύο-τρία χρόνια. Δεν είναι αγορά αυτή, είναι μια τεχνητή αγορά, πουλάμε τεχνητά αγαθά για να ικανοποιήσουμε κάποια ανάγκη ως αποτέλεσμα της πολιτικής Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μα πρέπει να μας καθοδηγεί αγορά και όχι τα φορολογικά συστήματα και συμφωνήσαμε πως θα πρέπει να είμαστε σε θέση να ρυθμίσουμε τα βάρη και η αγορά αντέδρασε ε, παρκώς. Και είναι προφανές πως ε, η παραγωγή στην Ευρώπη πέφτει Άρα υπάρχει λιγότερη ζήτηση για επενδύσεις. Οπότε η αγορά αντιδρά μέσω των τιμών με τρόπο επαρκή. Οι προθέσεις μας ήταν διαφορετικές, αλλά εάν ακολουθούσαμε τη λύση της αγοράς θα μπορούσαμε να μείνουμε σε αυτό. Εγώ έχω ακούσει μια έκθεση από την Deloitte για την αποτελεσματικότητα στα ζητήματα αυτά της παγκόσμιας οικονομίας και Οπότε λέει η Γερμανία η οποία είναι η μόνη ευρωπαϊκή χώρα η οποία θεωρείται υψηλή αποδοτικότητα κινδυνεύει να χάσει τη θέση της. Η Γερμανία η οποία είναι πάρα πολύ ανταγωνιστική. Υπάρχει πολύ υψηλό κόστος εργασίας και υψηλό κόστος ενέργειας στη Γερμανία. αν δεχτούμε λοιπόν την πρόταση της Κομισιόν η οποία θα έχει πάρα πολύ μεγάλες ε, συνέπειες, ε, θα καταστήσουμε τη γερμανική οικονομία αλλά και όλες τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές οικονομίες πιο δύναμες θα υποφέρουν από υψηλότερο κόστος ε, ενέργειας και θα χάσουν ανταγωνιστικότητα. Ευχαριστώ για δύο λεπτά τώρα. Οι υπόλοιποι συνάδελφοι. Μάρσιεβιτς. Ναι, ευχαριστώ. Ευχαριστώ πρόεδρε αυτή η αλλαγή σήμερα της οδηγίας όπως συζητείτε ουσιαστικά δίνει στην Επιτροπή μια εντολή απεριόριστη για την αλλαγή αυτού του δικαιώματος, παραγωγής δικαιωματών σύμφωνα με το 14 της οδηγίας. Θα πρέπει όλα αυτά να προβλέπονται σε σχέση με το ολοχρόνο διάγραμμα και πώς οργανώνται αυτοί οι διαγωνισμοί παραχώρησης και σχετικά και με τον όγκο των ποσοτήτων αυτών, κατόγκων. Εδώ οι παρεμβάσεις θα μπορούσαν να θεωρηθούν σαν πρόταση σταθερότητας για την αγορά και με την οδηγία, η οδηγία όμω είναι σε αντίθεση με το 290 άρθρο των συνθήκων και η παραχώρηση αυτή δεν μπορεί να αφορά τα κύρια σημεία της οδηγίας γιατί αυτά τα σημεία διέπονται από τη συναπόφαση. Και ακόμη, όσα προτείνονται επηρεάζουν τις δυνατότητες της αγοράς ουσιαστικά να αυτονομιμοποιηθεί, ας το πούμε έτσι, και η Επιτροπή με τις παρεμβάσεις της θα μπορούσε να δημιουργήσει μια αύξηση των τιμών που θα μπορούσε να επηρεάσουν αρνητικό τις ε, ε, επενδύσεις κυρίως στον τομέα παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος. Αυτές οι πρωτοβουλίες ε, της Επιτροπής δεν επηρεάζουν τις εκπομπές αλλά τις τιμές και μόνο. Και μέσω διαβουλεύσεων με τους πολίτες αποδείχτηκε ότι δεν δίνουν σημασία σε αυτές τις πρωτοβουλίες, γι' αυτό είμαστε κατά αυτών παρεμβάσεων. Η συνάδελφος Μποβίσκα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Η κυρία Χολ είπε πως είναι μια απλή πρόταση και πρέπει να το ευθύσουμε γρήγορα. Όμως, αυτός απλός κανονισμός ε, έχει οδηγήσει σε πολύ έντονη συζήτηση που θυμάμαι. Τη θυμάμαι εγώ από δεκαετία των 90 Πού είναι η λεπτή αυτή γραμμή μεταξύ αγοράς και σχεδιαζόμενης οικονομίας. Είναι μια συζήτηση που υπήρχε ήδη από δεκαετία του 80 και του 90, στην Πολωνία τουλάχιστον. Είναι ενδιαφέρουσα λοιπόν αυτή η συζήτηση. Ποια είναι η λεπτή γραμμή μεταξύ ε, σχεδιασμού της οικονομίας ε, και ρύθμισης αγοράς. Αυτό το οποίο συζητάμε τώρα είναι ένας φόρος άνθρακα που έχει μικρή σχέση με εκπομπές, ε, χρηματιστήρια κτλ. Από την πίσω πόρτα λοιπόν η Κομισιόν θέλει να περάσει αυτή την ιδέα του φόρου άνθρακα. Και αν η Κομισιόν μπορεί να ορίζει τις ε, τιμές ε, και τον αριθμό των αδειών κτλ. Τι είναι αυτό, μια ρύθμιση από την πίσω πόρτα. Ένα άλλο ζήτημα το οποίο με ανησυχεί είναι διαδικαστικό η Κομισιόν έχει ήδη αποφασίσει ποια θα είναι η μοίρα αυτού του θέματος και το Κοινοβούλιο απλά οφείλει να εγκρίνει τις ε, προτάσεις αυτές. Γιατί το έχουν πει ξεκάθαρα πως 900 εκατομμύρια άδειες θα αποσυρθούν από την αγορά. Και η Επίτροπος είπε σε μια ακρόαση της Επιτροπής Περιβάλλοντος πως πρέπει τώρα να υιοθετηθεί και από το Κοινοβούλιο. Εμείς δηλαδή μόνο για έγκριση είμαστε εδώ πέρα, μια συλλημένης απόφασης. Και το έχει πει πολλές φορές δηλαδή, τυπική έγκριση, αυτό είπε. Ίσως αυτό κατάλαβε η κυρία Χολ όταν λέει ε, πως ε, είναι πολύ απλή υπόθεση. Δεν είναι απλή η υπόθεση δεν είναι μια απλή ρύθμιση γιατί αυτό το πράγμα θα έχει συγκεκριμένα αποτελέσματα. και συνέπειες για βιομηχανίες ε, στην Ευρώπη κτλ. Οπότε τώρα τα λαμβάνουμε αυτά υπόψη όταν συζητάμε τέτοια ζητήματα. Σας ευχαριστώ. Βιντάλ Κόντρας. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε για την μεταρρύθμιση του καθεστώτος ε, της εμπορίας των δικαιωμάτων εκπομπών. Σίγουρα επηρεαζόμαστε από τις ιδιαίτερες συνθήκες που βιώνουμε αυτή την μακρά πολύ δύσκολη κρίση η οποία καταστρέφει και τον επιχειρηματικό ιστό, ιδίως ε, τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Μια κρίση που οδηγεί εκατομμύρια πολιτών στην απόγνωση και στην ανεργία. Η αύξηση των τιμών του άνθρακα έχει κάποιους στόχους, δηλαδή προσωρινή απόσταση των δικαιωμάτων εμπορίας και κατά την άποψή μου θα έχει ως αποτέλεσμα ε, και αύξηση των ε, τιμών ε, τη δραστηριότητα στην οποία σα περιέγραψα. Δηλαδή, αν τα προσθέσουμε αυτά στην κρίση, πολλέ επιχειρήσει εντατική χρήση ενέργεια θα επιλέξουν την μετεγκατάσταση και θα, χρειαστεί, θα χρειαστεί να καταβληθεί μεγαλύτερος λογαριασμός με μεγαλύτερη θυγό με την ανταγωνιστικότητα. Φυσικά καταλαβαίνετε ότι δεν μπορούσε να βρεθεί χειρότερη στιγμή για κάτι τέτοιο. Και από την άλλη πλευρά, κάτι που πάντα συμβαίνει. Όπως είπατε και εσείς, έχει ξεκινήσει η συνοδοκορυβή τη της Ντόχα. Είμαστε μέσω αυτή τη ε, διάσκεψη. Έχουμε ανταγωνιστέ που και αυτοί βέβαια εκπέμπουν πολύ μεγάλε ποσότητε διοξιδίου και φαίνεται ότι είναι και τόσο διατεθειμένοι να φτάσουν σε διεθνεί συμφωνίε και να συνεργαστούν μεταξύ του για να δημιουργηθεί ένα παγκόσμιο πλαίσιο αντιμετώπιση του προβλήματο. Επομένω, εμεί τι θα κάνουμε, θα συνεχίσουμε να πυροβολούμε το ίδιο μα το πόδι, ενώ οι άλλοι δεν κάνουν τίποτα. Αν θέλουμε, εντάξει, μπορούμε να το κάνουμε, αλλά δεν νομίζω ότι είναι και το πιο ευφιές. Και όπως παρακολουθούμε και τις εργασίες της διάσκεψης της Ντόχα, βλέπουμε ότι είναι και πολύ μικρές προσδοκίες. Το καθεστώς λοιπόν πληστηριασμού των δικαιωμάτων, όπως είπατε και εσείς πολύ σωστά, έχει τεχνητά δημιουργηθεί από πάνω προς τα κάτω. Άρα δεν είναι ε, με αυστηρένεια του όρου αγορά, όταν δηλαδή φυσικά και αυθόρμητα έχουμε από κάτω προς τα πάνω σαστικά τις συναλλαγές. Και έτσι δημιουργείται και αυτό το πρόβλημα που έχουμε αντιμετωπίσει αντιμετωπίσουμε σήμερα. Εάν λοιπόν δώσουμε στην Κομισιόν την εξουσία να παρεμβαίνει στις αγορές όταν το κρίνουμε αυτό ή το κρίνει ορθό, αυτό δεν ξέρω κατά πόσο να συμβατώ με την ασφάλεια δικαίου και την ίδια την έννοια της αγοράς. Εγώ θα έλεγα ότι δεν είναι. Οπότε η οδηγία, η οδηγία για την εμπορία των δικαιωμάτων υποβόλων και στο άρθρο 10 λέει ότι πρέπει να δυνατό να επιτρέπεται η ανάπτυξη της διαδικασίας ό,τι αφορά το χρονοδιάγραμμα με βάση το ρυθμό και με βάση τους όγκους ε, των δικαιωμάτων που τίθενται στη δάση κτλ. Τι θα κάνουμε λοιπόν όταν βλέπουμε εδώ να υπάρχει ουσιαστικά παραβίαση αυτής της διάταξης της οδηγίας. Υπάρχουν αντιφάσεις σίγουρα, αλλά όχι να τις κάνουμε μέθοδο εργασίας στις αντιφάσεις αυτές. Δεν νομίζω ότι είναι κάτι που μπορούμε να το υποστηρίξουμε. Μια στιγμή αφαιρέθηκα και ευτυχώς υποφελήθηκε ο συνάδελφος Βιντακουάντρας. Ρόι. Κυρία Πρόεδρε, αν δει κανείς την κατάσταση εδώ πέρα διαπιστώνει πως έχουμε χαμηλή ανάπτυξη οπότε χρειάζονται λιγότερα πιστοποιητικά επιχειρήσεις από ό,τι είχαμε υπολογίσει. Έχουμε υψηλότερη ενεργειακή αποτελεσματικότητα οπότε χρειάζεται, χρειάζονται λιγότερα δικαιώματα. Φτιάχνουμε περισσότερες ε, ΑΠΕ οπότε χρειαζόμαστε λιγότερα πιστοποιητικά. Μα αυτό θέλαμε. Απλά επειδή η κατάσταση τώρα στην οικονομία είναι διαφορετική από ό,τι θέλαμε και τα κράτη-μέλη δεν έχουν τα έσοδα που θέλανε, τι κάνουμε, ανεβάζουμε τις τιμές. Είναι αυθαιρεσία αυτό. Αποφασίσαμε αυτό το σύστημα γιατί θέλαμε ακριβώς ένα σύστημα αγοράς. Δεν μπορούμε όποτε δεν μας αρέσει να κάνουμε ό,τι θέλουμε. Δεν το καταλαβαίνω αυτό. λέτε πως δεν επιτυχαίνουμε τους όχους μας. Μα τους επιτέχουμε. Τους επιτυχάνουμε, με συγχωρείτε. Όλα συμβαίνουν εκτός από το ότι δεν υπάρχουν αρκετά έσοδα. Έμα ε, αυτό είναι λάθος προγραμματισμού των κρατών. Είναι δικό του πρόβλημα. Και δεν είναι τότε, α, θα τα ακριβίνουμε τα πράγματα. Είτε έχουμε ένα σύστημα αγοράς, είτε αυθαιρεσία. Αυτό το οποίο κάνουμε τώρα δεν προσφέρει ασφάλεια δικαίου, δεν προσφέρει σταθερότητα, είναι ακριβώς το αντίθετο ανοίγει την πόρτα για αυθαιρεσία και ο συνάδελφος Βιδάλ Κουάντρας έχει δίκιο. Είναι θεμελιώδης παρέμβαση αυτή η οποία συμβαίνει. Το σύστημα στο οποίο ε, βασιζόμασταν δεν ε, είναι σύστημα στο οποίο θα μπορούμε να βασιζόμαστε στο Δεν υπάρχει καμία ασφάλεια δικαίου. Τελείως λανθασμένο σύστημα. Και αυτά τα οποία σημαίνουν και στο κοινοβούλιο είναι σκανδαλώδη. Τα είπε η κυρία Κολάρ Σκαμπομίνσκα. Σκανδαλώδη οι πρόεδροι των μεγάλων ομάδων ε, παρακαλάνε τον πρόεδρο της ε, Κομισιόν να το ξαναδεί, δημιουργούνται εδώ πέρα τετελεσμένα. Είτε έχουμε δικαίωμα συναπόφαση ή δεν έχουμε. Ή κάνει η Κομισιόν ό,τι θέλει εκείνη. Αλλά αυτό δεν είναι δημοκρατία. Είναι και ουσιαστικά μπουρδα και είναι και περιφρόνηση του Κοινοβουλίου. Ευχαριστώ, Ντελκαστίγιο. Ναι, ναι, ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Σε αυτή τη μικρή δικαιολογία της διαδικασίας ε, αυτό ότι δεν θα μειωτεθεί μέσω και της επιτροπολογίας, έστω για λογικό ε, ελπίζει αυτό από το Κοινοβούλιο και την αλλαγή του 10 παράγραφος 4 άρθρου ούτε την βοήθεια ή όχι των όσων γίνονται στην αγορά, αλλά ποια είναι η αχίλιος πτέρνα της σχετικής πρότασης. Είναι το εξής. Εκεί που αλλάζουν τα πράγματα για ίσες ευκαιρίες για όλους για να μπορούσαν να ανταγωνιστούν μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχουμε την εξή ε, λογική ανάλυση. Αν δεν έχουμε πια δικαιώματα 900 εκατομμύρια τόνους για εκπομπές ε, αυξάνεται η τιμή του άνθρακος. Και όπως συμβαίνει από το 2013 και μετά, τι έγινε. Ίσως υπάρξουν άμεσες ενισχύσεις στις βιομηχανίες που καταναλώνουν πολλή ενέργεια, εντατικά μάλιστα, και μόνο στα κράτη εκείνα που μπορούν να χορηγήσουν αυτή την άμεση ενίσχυση, τότε καταλαβαίνετε ότι έτσι θα υπάρξει αυτό η ανταγωνιστικότητα από αυτέ. Θα αυξηθεί η τιμή, αλλά ταυτόχρονα εάν δεν υπάρξουν άμεσε ενισχύσει σε, σε αυτά τα εργοστάσια, αλλά τα κράτη, διάφορα κράτη-μέλη να μπορούν τα ίδια να δίνουν αυτά τα πράγματα, τότε υπάρχουν ανισότητες που δημιουργούνται Καταλαβαίνετε το νόημα, για τις συνθήκες αυτές, για ίσο ανταγωνισμό, σωστό ανταγωνισμολογικό. Να, τα κράτη-μέλη να μην μπορούν να δίνουν ε, άμεσες ενισχύσεις ε, σε αυτές αυτά τα εργοστάσια είτε να υπάρξει μια εναρμόνιση της όλης νομοθεσίας ε, και σε όλα τα κράτη-μέλη να μπορούν να χορηγούν Εντάξει, ή το ένα να ισχύσει το άλλο. Διαφορετικά δεν γίνεται. Δεν μπορούμε να προχωρήσουμε. Αυτή είναι το αδύναμο σημείο και δεν υπάρχουν πια οι ιδανικές συνθήκες ανταγωνισμού της βιομηχανίας στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε και να πω πόσο ικανοποιητικό είναι που συμφωνώ με τους περισσότερους συναδέλφους που ήδη μίλησαν και τον κύριο Ρόλ και τον κύριο Βιδάλ Κουάντρας που επέμειναν πως το ETS ε δεν είναι ε, σωστός μηχανισμός αγοράς. Εγώ αυτό το λέω εδώ και 2-3 χρόνια. Είναι ένας τελείως τεχνητός και γραφειοκρατικός μηχανισμός. Αφορά κάτι το εικονικό και όχι πραγματικό και είναι, θα έλεγα, αποτέλεσμα γραφειοκρατικής διαταγής και είναι άρα αδύνατον να προγραμματίσουν οι επιχειρήσεις. Τώρα βλέπουμε πως οι προβλέψεις αυτές ήταν σωστές, δεν υπάρχει βεβαιότητα. Η Κομισιόν θεωρεί πως μπορεί να παρεμένει και να αλλάζει τους όρους όποτε θεωρεί ότι κάτι τέτοιο χρειάζεται και το έκανε και πάλι. Εγώ λέω πως εάν πρέπει να υπάρξει ένα αντικίνητρο τότε με οικονομικούς όρους ένας φόρος, αν και δεν μου αρέσουν οι φόροι, θα ήταν πολύ πιο αποτελεσματικός. Και τώρα στη χώρα μου το Ηνωμένο Βασίλειο έχουμε τον Υπουργό Οικονομικών που θα θέσει μάλιστα κατώτατο όριο της τιμής του άνθρακα για να ξεπεράσει τις ξεκάθαρες αποτυχίες του συστήματος. Και πρέπει να πούμε πως τη ΣΥΠΑ οι εκπομπές μειώνονται όχι λόγω κάποιων φοβερών γραφειοκρατικών μηχανισμών, αλλά ως αποτέλεσμα των δυνάμεων της αγοράς. Αυτό είναι μάθημα για όλους μας, μάθημα για την Ευρώπη και καλά θα κάνουμε να το σημειώσουμε. Ειδικά σε καιρό που πολλοί μεγάλες ποσότητες ε, αερίου σε σχιστόλιθο φαίνεται πως ανακαλύπτονται στην Ευρώπη. Ευχαριστώ Ρουμπίχ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Θεωρώ πως αυτό το οποίο διαπιστώνουμε τώρα, το είδαμε και στις ειδήσει, είναι πως κλείνουν χαλιβουργίες στην Ιταλία και στην Ισπανία. Ένα τρίτο της παραγωγής, ε, λέει η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία, πως πρέπει να κλείσει γιατί δεν είναι ανταγωνιστική η Ευρώπη. Και τώρα η Κομισιόν λέει πως μέχρι το 20% ε, του ΑΕΠ θα πρέπει να πάει στην επαναβιομηχάνηση. Μα με την πολιτική που ακολουθούμε, δηλαδή δεν στηρίζουμε τις επιχειρήσεις που κινδυνεύουν να φύγουν, αλλά θέλουμε να τις επιβαρύνουμε, πώς θα δημιουργήσουμε νέες θέσεις εργασίας στη βιομηχανία. Χάνονται δεκάδες χιλιάδες θέσεις εργασίας και τι θα κάνουμε, δηλαδή κρατικοποίηση όπως λέει τώρα η Γαλλία, δεν θα επιτύχουμε έτσι τους ε, στόχους μας. Ε, λαμβάνει χώρα διάσκεψη στην Ντόχα, όσοι θα πάνε εκεί ε, πετώντας να κοιτάξουν εκεί πέρα το εργοστάσιο αλουμινίου που μετακόμισε από την ε, Νορβηγία στην Τόχα γιατί είναι πολύ πιο φτηνές οι τιμές του αερίου. Πρέπει να δούμε λοιπόν πώς θα κρατήσουμε τις μεγάλες αυτές επιχειρήσεις ε, στην Ευρώπη πώς θα διαμορφώσουμε το σύστημα αυτό για να εγκατασταθούν εδώ πέρα οι καθαρότερες επιχειρήσεις του κόσμου. Όχι να στέλνουμε τις επιχειρήσεις μας στην Αμερική να μην τηρούν εκεί πέρα τις ε, διατάξεις, να ρηπαίνουν το περιβάλλον και εδώ πέρα να χάνουμε θέσεις εργασίας. Δεν είναι δυνατόν. Θεωρώ πως σωστή απάντηση είναι να μην ε, φορολογούμε τις ε, επιχειρήσεις που ανταγωνίζονται διεθνώς, γιατί οι Κινέζοι, οι δεν έχουν τέτοιους φόρους. Πρέπει να προτείνουμε έναν φόρο ε, στα προϊόντα ε, ένα 2-3% παραπάνω στο ΦΠΑ αναλόγως με το που παράγονται και από που προέρχονται. Το σύστημα του ε, ETS είναι λανθασμένο, προκαλεί ανεργία στην Ευρώπη και δεν μπορούμε να το επιτρέψουμε αυτό. Ευχαριστώ Μπρεζίνα. Ευχαριστώ. Κυρίες και κύριοι, κυρία Πρόεδρε, εγώ θυμάμαι μια εποχή όταν ε, πολλοί από εσά ε, υπερψήφιζαν ε, το ETS. Και οι βουλευτές εκείνοι που είχαν υπερψηφίσει μας λέγανε πως μπορεί να είναι γραφειοκρατικός ο μηχανισμός αλλά βασίζεται σε κάποιες αρχές της αγοράς. Εγώ είχα καταψηφίσει τότε mm-hmm. και νομίζω πως τώρα είναι η στιγμή να ξυπνήσουμε και να σταματήσουμε να το κάνουμε ακόμη πιο περίπλοκο από όσο είναι. Επίσης θεωρώ πως ε, αντί να επενδύουμε σε αυτό το σύστημα πρέπει οι επενδύσεις αυτές να πάνε σε νέες τεχνολογίες πιο πράσινες όπως κάνουν οι ΙΠΑ. Μόλις ακούσαμε πως οι εκπομπές εκεί πέρα έχουν μειωθεί σημαντικά. Εγώ θεωρώ πως πρέπει να καταψηφίσουμε αυτή την πρόταση. Αλλά επίσης θεωρώ πως τώρα έχει φτάσει η στιγμή να ξανασκεφτούμε τη γενικότερη προσέγγιση μας ε, στο ζήτημα αυτό. Και ίσως να καταλήξουμε σε κάτι καινούργιο δεδομένη της οικονομική κρίση. Ευχαριστώ. Συνάστος πρώτη. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Ορισμένες αφιβολίες έχω εγώ. Το ETS ε είναι μηχανισμός της αγοράς. Δυσκολεύομαι ξεκινώ να καταλάβω. Μηχανισμός αγοράς όπου περίπου το 50% των εκπομπών δωρεάν παραχωρείται. Μια αγορά δεν μπορεί να λειτουργεί κατά από αυτές τις συνθήκες. Πάντως, μέσα σε αυτή την οικονομική κρίση, πέρα από την αγορά αερίου στις ΗΠΑ Πολιτείες, αλλά και στα υπόλοιπα ορυκτά καύσιμα εδώ, πραγματικά νιώθει την αγορά και νιώθει την κρίση και έχουμε μια αλλαγή των τιμών. Το σημερινό επίπεδο κόστους για δικαιώματα εκπομπής ουσιαστικά είναι το κόστος αυτό πολύ, χαμηλά, πολύ χαμηλό σε σχέση με τις δυνατότητες της αγοράς, τις ποσότητες στην αγορά. Εμείς λοιπόν δεν νομίζω ότι μπορούμε έτσι να ενεργούμε στην αγορά αυτή. Εάν ε, η πρόθεσή μας δεν είναι πραγματικά σοβαρή σε γενικό επίπεδο να υιοθετήσουμε το πρωτόκολλο του Κιώτο. Εάν είναι το, πρώτο, το πρωταρχικό μας σχέδιο για μας, δεν γίνεται. Πρέπει να έχουμε και μια αναλλακτική λύση, ένα σχέδιο Β. Ποιο είναι? Να έχουμε ένα τέλος αντιθαθμιστικό στα σύνορα. Η Άσα προϊόντα προέρχονται από χώρες που δεν είναι πειθαρχημένες ε, στην εκπομπή αερίων με φαινόμενο θερμοκηπίου. Ευχαριστούμε τον αδελφό πρώτη. Οντί. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε για να πω και εγώ κάποια σχόλια μετά από τα διαφωτιστικά σχόλια των συναδέλφων. Διαρωτώ με μήπως τελικά πετάμε μαζί με τα ξέρα και τα χλωρά γιατί τι εντύπωση έχω αποκομίσει, κυρία Πρόεδρε. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα έπρεπε να είχε κάνει μια αξιολόγηση αυτού του μηχανισμού, αυτού του συστήματο. Πιστεύω ότι αυτό το σύστημα ήταν καινοτόμο. Ότι βρισκόμαστε στη φάση, αν θέλετε, του πολιτικού πειραματισμού ενό πάρα πολύ σημαντικού πολιτικού στόχου που είναι ο περιορισμό ε, των ποσοστώσεων ε, των εκπομπών μα. Με πλαίσιο, το, μάλλον με ορίζοντα το 2020 και με ποσοστό 20%. Δεν ξέρω αν θα έπρεπε να γίνει μια αξιολόγηση για να δούμε ακριβώ πώς λειτουργεί αυτός ο μηχανισμός. Τα κράτη-μέλη κάνουν την κατανομή, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επιβλέπει και τώρα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή Μα ζητά με μία σελίδα να της δώσουμε σημαντικές εξουσίες και τελικά να προσαρμοστεί η λειτουργία της αγοράς. Εμείς οι βουλευτές μπορούμε όμως να αποφασίσουμε ότι αντίθετα θα θέλαμε μία αρχή ε, υπεύθυνη για αυτήν την αγορά όπως ψηφίσαμε σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά μια πολιτική ε, αρχή ευρύτερη, μια πολιτική εξουσία δηλαδή για να δούμε αν αυτό το οποίο έχουμε δημιουργήσει πρώτον λειτουργεί σωστά, δεύτερον τι θέλουμε να κάνει και τρίτον έχουμε και μια πραγματική αξιολόγηση. Το άρθρο 25 για παράδειγμα προβλέπει ότι θα πρέπει να συναυτούν συμφωνίες με τρίτες χώρες που είναι συμβαλόμενα μέρη του πρωτοκόλλου του Κιώτο. Αυτό προβλέπεται. Έχουν συναυτεί συμφωνίες. Ποιε σχέσεις διατηρούμε με άλλες περιοχές του κόσμου σε σχέση με αυτό το πειραματισμό, αν θέλετε. Γίνονται αντίστοιχα πειράματα άλλου στον κόσμο υπάρχει και ένα εντελώ διαφορετικό πρόβλημα. Αυτό ο φόρο για τον άνθρωπο, για παράδειγμα. Αυτό είναι τελείω διαφορετικό. Εδώ ε, μιλάμε για τι εκπομπέ ε, των εισαγωγών ε, και το άλλο αφορά το φόρο του άνθρακα. Είναι διαφορετικά πράγματα. Εγώ λοιπόν θα ήμουν υπέρ του να γίνει μια πραγματική αξιολόγηση γιατί αυτό θα μα δώσει τη δυνατότητα να συζητήσουμε και στο πλαίσιο προεκλογική εκστρατεία για τι ευρωεκλογέ του 2014, να έχουμε μια πραγματική πολιτική συζήτηση απέναντι στους συμπολίτε μας για το σύνολο του όλου μηχανισμού. Πολύ καλά. Η Επιτροπή η Ευρωπαϊκή έχει το λόγο τώρα. Ποιος παρίσταται. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ακούσαμε με μεγάλο ενδιαφέρον τις παρεμβάσεις των βουλευτών. Θα ήθελα να αναφερθώ σε κάποια πράγματα. Πρώτα απ' όλα την κατάσταση η Κομισιόν ανέλησε την ε, κατάσταση. Τον Ιούλιο είχαμε ένα έγγραφο που ανέλυε την κατάσταση, σας το δώσαμε και πριν από δύο εβδομάδες βγάλαμε μια αξιολόγηση αντικτύπου που κοιτάει την ε, σημερινή αγορά σε βαθμό λεπτομέρειας και βεβαίως λέμε να αλλάξουμε τους ε, Πληστηριασμού ε, και να βγουν εκτός 900 εκατομμύρια άδειες. Έχει γίνει λοιπόν τεχνική ανάλυση και από τη διαβούλευση με τους ενδιαφερομένους που κάναμε το καλοκαίρι νομίζω πως το αμφισβητεί κανείς πως υπάρχει αυτή τη στιγμή υπερβολική παροχή αδειών στην αγορά. Αυτό προκαλείται από την οικονομική κρίση, από την άλλη από ρυθμιστικές αποφάσεις που λήφθησαν στο επίπεδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από τα κρατη και από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο όταν μιλάμε για κάποιες ε, άδειες οι οποίες δόθηκαν και σε ανσόμενες χώρες. Ε, έχουμε λοιπόν μια ανισορροπία που θα πρέπει να προσπαθήσουν να αντιμετωπίσουν και οι εταιρείε, δηλαδή εάν δεν υπάρχει αρκετή, αν δεν υπάρχει αρκετή ζήτηση η εταιρεία θα αποσύρει κάποια δικαιώματα και το ίδιο κάνουμε και εδώ πέρα. Δεν νομίζω να κάνουμε τίποτα το εξαιρετικό. Αυτό το οποίο επίσης κοιτάμε και πρέπει να λάβουμε υπόψη είναι πως αυτά είναι περιουσιακά στοιχεία των κρατών μελών. Είναι φυσιολογικό ε, τα κράτη-μέλη να συνεχίσουν να βγάζουν τέτοια πράγματα στην αγορά όταν η τιμή είναι αυτή η οποία είναι. Δεν είναι λοιπόν κεντρικά σχεδιαζόμενη οικονομία, απλά κοιτάμε να δούμε ποιε ποσότητε θα διαθέσουμε και πότε. Επίση πρέπει να λάβουμε υπόψη πω αυτό δεν επηρεάζει καθόλου το συνολικό ποσό αδειών που θα είναι διαθέσιμε στη φάση 3, δηλαδή μεταξύ 2013 και 2020. Οπότε δεν είναι αυτό το οποίο προτείνουμε να κάνουμε μέσω της επιτροπολογίας που είναι όντως η πράξη κατεξιοδότηση. Αυτό το οποίο προτείνεται στο Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο μέσω τη ακτική νομοθετική διαδικασία είναι να ξεκαθαρίσουμε την νομική εντολή ότι κάτι τέτοιο μπορεί να γίνει και αυτό βέβαια έχουμε υποβάλει σε εσάς. Και στις 25 Νοεμβρίου επίσης ε, είπαμε πως ε, δεν σκοπεύουμε να κρίνουμε βέβαια σε αυτά τα οποία έχει οφθεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Εμείς δεν θα υιοθετήσουμε τυχόν τέτοιες ε, ε, προτάσεις, τις προτάσεις που έχουμε κάνει δηλαδή, μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία λήψη αποφάσεων ε, εντός του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. Οπότε δεν προδικάζουμε τίποτα. Τώρα, πράγματι η Κομισιόν ε, έχει κάνει αυτή την πρόταση για την απόσυρση 90, 900 με συγχωρείτε, εκατομμυρίων τέτοιων αδειών, αλλά βεβαίω αυτό θα το εξετάσει το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο επί τρει μήνε. Οπότε δεν προδικάζουμε τίποτα αναφέρθηκε πως θα πρέπει να κοιτάμε μόνο τα διαρθρωτικά μέτρα πως όλα αυτά καλά είναι αλλά πρέπει να δούμε τι πρέπει να γίνει από διαρθρωτική πλευρά για να φτάσουμε σε αυτή την οικονομία χαμηλού άνθρακα που θέλουμε όλοι Και βέβαια εκεί πέρα έχουμε κάποιε επιλογέ για διαρθρωτικά μέτρα που μπορούν να ληφθούν για την ενίσχυση του συστήματο εμπορία εκπομπών. τέλο. η πρόταση αυτή τη απόσυρση είναι τεχνική για να αποφύγουμε την κινητικότητα γιατί αυτή τη στιγμή υπάρχει πάρα πολύ χαμηλή τιμή. Αριθμίσουμε λοιπόν τώρα λίγο την ε, προσφορά. Μπορούμε να έχουμε πολύ πιο σταθερές τιμές και έτσι οι τιμές δεν θα έχουν ψεύτικες προσδοκίες, δηλαδή να έχουν χαμηλέ τιμές αύριε. σήμερα και αύριο υψηλέ αυξήσει. Τέλος, έγινε μια αναφορά σε τρίτες χώρες, ε, τη διάσκεψη τη Ντόχα η οποία ξεκίνησε. Να αναφέρω πως πράγματι είχαμε πάρα πολύ καλές επαφές με τρίτες ε, χώρες. Γνωρίζετε πως ήδη υπάρχει σύνδεση μεταξύ του συστήματος αυτού και του συστήματος της Αυστραλίας. Τότε εργαζόμαστε από αυτού. Είχαμε πάρα πολύ καλές επαφές επίσης με την Κίνα για πιλωτικά έργα και θα ήταν πάρα πολύ κρίμα εάν η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορεί να δείξει πως ε, το σύστημα το οποίο έχει επηρεαστεί από την οικονομική κρίση δεν ε, μπορούμε να το διατηρήσουμε. Και θα είναι μια χαμένη ευκαιρία για να πείσουμε και τις άλλες ε, χώρες να λάβουν σοβαρά τέτοια μέτρα. Δείχνοντα λοιπόν πως μπορούμε να διατηρήσουμε το σύστημα αυτό με λογικέ τιμές και όχι παράλογες τιμές, παράλογα χαμηλέ. ελπίζουμε πως το Κοινοβούλιο θα δει τις προτάσει αυτέ θετικά. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Για να ακούσουμε τώρα και από πλευρά εισηγητού τι γίνεται. Εγώ πιστεύω ότι ολοκληρώσαμε τη διαδικασία αυτή με επιτυχία. Δηλαδή αυτή ήταν ανταλλαγή απόψεων, ήταν μια πραγματική ανταλλαγή απόψεων. Ακούσαμε και διαφορετικές απόψεις, διαφορετικές από, αυτή, από αυτές του βέβαια. Ο εισηγητής σας θα ήθελε να ακούσει περισσότερους να συμφωνούν με τη δική του θέση. Αλλά έτσι έχει αυτή η διαδικασία. Αποτελεί τμήμα της εξέτασης αυτής της νομοδότησης και θα δούμε πώς θα εξελιχθούν οι απόψεις των ε, διαφόρων πολιτικών ομάδων και πώς επίσης θα εξελιχθεί και το έγγραφο το οποίο θα εκπονήσω ως εισηγητή σας. Πρέπει να υπενθυμίσω ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ζήτησε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να δεσμευθεί ότι θα αλλάξει τον, ε, το χρονοδιάγραμμα πληστηριασμών στο πλαίσιο της οδηγίας για την ενεργειακή απόδοση. Δεν μπορούμε τη μία να εγκρίνουμε κάτι και την επόμενη μέρα να το ξεχνάμε και να ζητάμε κάτι διαφορετικό. Επομένω, νομίζω θα πρέπει τουλάχιστον να επιδεικνύουμε κάποια συνέπεια ε, στο νομοθετικό μα έργο ως Κοινοβούλιο. Είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να αποτελεί στόχο. Θα ήθελα να επιμείνω στη θέση την οποία σας ε, ξέθεσα στην αρχή. Όπως είπα, είμαι υπέρ της πρότασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, απλά θέλω να διευκρινίσω και να προσθέσω και το εξή. Είναι λογικό ότι η δική μου θέση και τοποθέτηση θα συμπληρωθεί με την ιδέα ότι η εξουσία που εκχωρείται στην Κομισιόν είναι προσωρινή και έκτακτη. Δηλαδή δεν μπορεί να αποτελέσει μια τακτική μόνιμη εξουσία, γιατί αυτό θα άλλαζε τελείως τα δεδομένα στην αγορά. Άρα είναι κάτι ε, που θα ισχύσει προσωρινά και έκτακτα. Δεν θα πρέπει λοιπόν να χαλαρώσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Πρέπει να εξακολουθήσει να σκέφτεται με ποιο τρόπο μπορεί να διατηρήσει ζωντανή αυτή την αγορά. Γιατί η αγορά αυτή, αν είναι ζωντανή, πραγματικά ανταποκρίνεται στις απαιτήσει και στις πολιτικές που έχουν εγκρίνει ελεύθερα εκούσια οι διάφορε τοπικέ αρχέ, προστάσεω περιβάλλοντο, μηχανική πολιτική κτλ. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει λοιπόν να εξακολουθήσει να εργάζεται προ αυτήν την κατεύθυνση, ώστε η αγορά αυτή να παραμείνει ζωντανή και να αποδώσει και στη συνέχεια του καρπού που αποδίδει μέχρι στιγμή. Ευχαριστώ. Σα ευχαριστώ πολύ. Ολοκληρώνεται λοιπόν η συζήτηση για το σημείο αυτό. Ακριβώ για τι 17 Δεκεμβρίου έχουμε προθεσμία, έχουμε τροπολογία. Μάλλον μέχρι την η 18 το μεσημέρι είναι η προθεσμία, έτσι. Να περάσουμε στο επόμενο σημείο της ημερησίας διάταξης. Ποιο είναι αυτό? Σον Κέλλη. Ελεύθερη κυκλοφορία ατόμων. Σον Κέλλη. δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Πρόεδρε. Χαίρομαι ιδιαίτερα παρουσιάζω την έκθεσή μου. Ευχαριστώ. Μισό λεπτό να περιμένουμε να αποχωρήσουν Παρακαλώ, σε επιθυμούν να αποχωρήσουν, να το κάνουν τάχιστα για να μπορέσουμε να συνεχίσουμε. Uh, Ευχαριστώ. Χαίρομαι που παρουσιάζω το σχέδιο έκθεσης για τον κανονισμό προστασίας προσωπικών δεδομένων. Και να πω πως αυτή τη στιγμή είχα μέχρι αυτή τη στιγμή είχα πάνω από 100 συναντήσεις με επιχειρηματίες ΜΚΟ ενδιαφερομένους και υπάρχει πολλή δουλειά που πρέπει να γίνει και ενδιαφέρει πάρα πολύ τον κόσμο ειδικά όσον αφορά την ε, επικαιροποίηση της οδηγίας του 1995 για την εποχή των κοινωνικών δικτύων του ηλεκτρονικού εμπορίου είναι μια μεγάλη πρόκληση. Η Κομισιόν έχει μια φιλόδοξη προσέγγιση και πρέπει να την επενέσουμε και επίσης βεβαίως πρέπει να εφαρμόσουμε και το άρθρο 8 της Χάρτας Θεμελιωδών Δικαιωμάτων ε, αφού πέρασε η συνθήκη της Λισαβόνας. Επίσης θα ήθελα να τονίσω τα, την πτυχή εσωτερικής αγοράς. Το άρθρο 114 παράγραφος 1 της συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, τα αναφέρει αυτά μαζί με το άρθρο 16. Εμείς λοιπόν στην Επιτροπή μας έχουμε να παίξουμε ένα ρόλο κλειδί στη διαμόρφωση αυτού του κανονισμού για να διασφαλίσουμε πως ο συμπεφωνημένος στόχος για τον υψηλότερο βαθμό προστασίας των προσωπικών δεδομένων δεν οδηγεί σε κάποιες ε, συνέπειες οι οποίες θα είναι η υπερβολική γραφειοκρατία. Και αυτό είναι ένας φόβος υπαρκτός. Επίσης, πρέπει να απλοποιηθούν οι κανόνες ε, για να υπάρξει καινοτομία, να μειωθεί το διοικητικό βάρος και να δημιουργήσουμε ένα περιβάλλον όπου δεν θα μπορεί να ε, ανθίσει καμία επιχείρηση και καμία ιδέα. Η εμπιστοσύνη είναι αυτό το οποίο έχουμε χρησιμοποιήσει πιο συχνά σχέση με αυτόν τον κόσμο Πρέπει επίσης ε, τα νέα προϊόντα και υπηρεσίες να έχουν την εμπιστοσύνη των πολιτών για να προωθήσουμε την καινοτομία και τη δημιουργικότητα ως εισηγητή, η δική μου προτεραιότητα είναι να διασφαλίσω πω το τελικό κείμενο θα περιέχει ε, την σωστή ισορροπία μεταξύ θεμελιωδών δικαιωμάτων και την ανάγκη ίσων όρων ανταγωνισμού και καινοτομία ε, των ε, εταιριών. Θα πρέπει λοιπόν να υπάρχει η δυνατότητα οι εταιρείε να απευθυνθούν σε μία και μόνη υπηρεσία. Περνάω τώρα σε κάποιες από τις βασικές πτυχές της εκθεσής μου. Μέτρα εταιρική διακυβέρνησης, τα οποία θα βασίζονται στην αρχή της λογοδοσίας, μια ποσοτική αντί για ποιοτική ε, προσέγγιση, η συνένεση ως βάση της επεξεργασίας, αλλά όχι ιδιαίτερη έμφαση σε αυτήν, να διατηρηθεί η εξαίρεση για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και οι διατάξεις εκείνες οι οποίες θα προωθήσουν τον ανταγωνισμό. Έχω προτείνει συνολικά 164 τροπολογίες στην πρόταση της Κομισιόν προτινόμενες αλλαγές. Θα πρέπει να μειώσουν το υπερβολικό διοικητικό βάρος για τις επιχειρήσεις, ειδικά τις επιχειρήσεις εκείνες οι οποίες έχουν ήδη ενσωματώσει τέτοια στοιχεία και εγγυώνται και ένα βαθμό ευελιξίας ειδικά αυτές που αφορούν τους μηχανισμούς λογοδοσίας. Κάποιοι ορισμοί και πτυχές του αρχικού κειμένου επίσης πρέπει να ξεκαθαρίσουν, να μπουν σε ένα νέο πλαίσιο και να απλοποιηθούν. Έχω λοιπόν προτείνει μια ποσοτική και όχι ποιοτική προσέγγιση η οποία θα βασίζεται στην εταιρική διακυβέρνηση που θα βασίζεται στη λογοδοσία όπως ανέφερα και όχι ε, ιδιαίτερη έμφαση στην ε, συνένεση, μια γραφειοκρατική διαδικασία, η οποία παρόλα αυτά έχει τη θέση της και αυτή. Σημαντικό είναι να δώσουμε επίσης έμφαση στον ρόλο τεχνικών λύσεων, όπως η ανωνυμοποίηση των δεδομένων από τον σχεδιασμό ήδη, καθώς επίσης και στοχευμένα μέτρα συμμόρφωσης. Όσον αφορά τώρα τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, έχω ζητήσει από τη μονάδα αξιολόγηση αντικτύπου του Κοινοβουλίου να κάνει μια αξιολόγηση η οποία θα παρουσιαστεί στην επόμενη συνεδρίαση της Επιτροπής μας 17 ε, Δεκεμβρίου, στις 7 με συγχωρείτε, Δεκεμβρίου. Ζητάω λοιπόν από τους συναδέλφους να στηρίξουν αυτή τη διάταξη. Επίσης έχουμε και τη φορητότητα των δεδομένων. Θεωρώ πως θα πρέπει να έχουμε ένα πλαίσιο το οποίο θα είναι τεχνικά εφικτό για να προσφέρει στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις ε, εναλλακτικές λύσεις όταν θα ε, αγοράζουν λύσεις δικτύου. Θεωρώ λοιπόν πως ε, το να διατηρήσουμε το άρθρο 15 θα είναι φιλικό για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Επίσης προσπάθησα να απλοποιήσω τις ε, διαδικασίες καταγραφής. Θεωρώ πως οι υπερβολικές τέτοιες διαδικασίες είναι γραφειοκρατικές και θα αφιερωθούν οι πόροι σε μέτρα ποσοτικά και όχι ποιοτικά. Επίσης, η πρώτερη αδειοδότηση θα είναι δύσκολη. Οπότε το έχω ξεκαθαρίσει αυτό ζητώντας μια πρώτερη διαβούλευση με τις αρχές προστασίας προσωπικών δεδομένων. Επίσης, οι ειδοποιήσεις για παραβιάσεις και οι κυρώσεις έχουν γίνει πιο πρακτικές στο σχέδιο εκθεσίσμου. μου. Ας δούμε λοιπόν τις πιθανώς ε, βλαβερές τέτοιες παραβιάσεις και να ενημερώνουμε τους ανθρώπους μόνο όταν απειλούνται υπό τρόπον ποιοτικό. Επίσης πρέπει να υπάρχει ελευθερία τύπου, κάτι το οποίο σκοπεύω να κάνω με τις τροπολογίες 1 και 154 όσον αφορά τα ερευνητικά τμήματα αυτά. Έχω εστιάσει στην έρευνα της υγείας. Έχω κάνει και ένα σεμινάριο. Η τροπολογία μου 9 για την ευρεία συνένεση και η τροπολογία 19 στόχο έχουν να δουν τις πιθανές ε, μη εσκεμμένες ε, συνέπειες. Επίσης ε, σκοπεύουμε να καταπολεμήσουμε το οικονομικό έγκλημα στην τροπολογία 28 και τον νέο άρθρο 23α. Επίσης η απάτη στον αθλητισμό είναι ιδιαίτερα σημαντική αν σκεφτούμε τα σκάνδαλα του ντόπινγκ, γι' αυτό έχω υποβάλει και τις τροπολογίες 70 και 71. Θέλετε να επιταχύνω? Ωραία. Ένα βασικό ζήτημα για την Επιτροπή μας είναι βεβαίω και η ενεργειακή αποτελεσματικότητα, γι' αυτό σκοπεύω να ε, υπάρξει κάποιο περιθώριο για έξυπνα δίκτυα στις, ε, στην τροπολογία 32 στο άρθρο 6 παράγραφος 4. Ε, θα προχωρήσω γρήγορα γιατί θέλετε να προχωρήσω γρήγορα θα πέρασε κάποια άλλα σημεία. Άρθρο 6 παράγραφος 4 ορίζει πως βάση για νόμιμη επεξεργασία δεδομένων ε, τα οποία δεν είχαν αρκετά συλληφθεί για αυτό το σκοπό αποτελεί ο έλεγχος των ενδιαφερομένων. Εγώ ήμουν κάπως προκλητικός με αυτή την τροπολογία γιατί θέλω να ξεκινήσει μια συζήτηση για το τι σημαίνει ακριβώς το θεμητό και νόμο ενδιαφέρον των ελεγκτών χωρίς να κινδυνεύσει η ιδιωτικότητα. Και να κινδυνεύσουν ε, νόμιμοι οικονομικοί τομείς. Τέλος, έχω εξετάσει μακρόν το πώς μπορεί να απλοποιηθεί η σχέση μεταξύ του υποκειμένου και του ελεγκτή ή αυτού ο οποίος επεξεργάζεται τα δεδομένα. Αυτή ορίζεται στο άρθρο 96 και περιέχει κάποιες μη συνέπειες που σημαίνουν πως αντί για μείωση των δεδομένων μπορεί αυτοί οι οποίοι εξεργάζονται τα δεδομένα να γίνουν έλεγκτες και να έχουν άμεση σχέση με τα υποκείμενα. Αυτό, κατά την άποψή μου, η σχέση αυτή πρέπει να διέπεται από το δίκαιο των συμβάσεων με βάση κάποια υποδείγματα σύμβασης. Θα πρέπει να απευθύνονται σε ένα σημείο βεβαίω οι ενδιαφερόμενοι και θα πρέπει να ασχολούνται με λοιπούς ανθρώπους. Δηλαδή, αν αγοράσει κανείς ένα αυτοκίνητο με εγγύηση, να πηγαίνει στον αντιπρόσωπο που το αγόρασε, όχι στο εργοστάσιο όπου φτιάχτηκε. Αναμένω λοιπόν και την αντίδραση των συναδέλφων επ' αυτού. Τέλος, ευχαριστήσω λοιπόν τον ε, Γιάννα Άλμπρεχτ ε, και του υπόλοιπους και οδησηγητές, δηλαδή τον Άξελφος και τους συνεισηγητές μου στην Γιούρη, ΙΜΚΟ και την Επιτροπή Περιβάλλοντος. Και έχουμε κάνει πάρα πολλή δουλειά τους τελευταίους ε, εννέα μήνες και θα συνεχίσουμε να το κάνουμε. Ευχαριστώ. Συγγνώμη, σας παρότρινα να ολοκληρώσετε, αλλά περνάει η ώρα και για παρακαλώ και οι σκιώδεις συγκητές που σε λίγο θα πάρουν το λόγο, αν είναι δυνατόν να περιοριστούν στα τρία λεπτά λόγο. κάου έχει το λόγο. Ευχαριστώ. Θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο Κέλλη με τον τρόπο με τον οποίο παρουσίασε τη γνωμοδότηση αυτή και πρέπει να σας πω ότι μέχρι ενός βαθμού μπορούμε να υποστηρίξουμε την προσέγγιση του. Δυστυχώς όμως υπάρχουν πολλές περιπτώσεις που οι τροπολογίες αποδυναμώνουν την αρχική πρόταση. Θα ήθελα να αναφερθώ εδώ στην επιτροπολογία, για παράδειγμα. Από αυτή την πλευρά, εμείς συμφωνούμε με τον εισηγητή κύριο Κέλλη, ότι δηλαδή η κατεξουσιοδότηση πράξη και οι εκτελεστικές πράξεις πρέπει να είναι περιορισμένες για να μπορούμε να διατηρούμε μια τεχνολογική ουδετερότητα. Θα θέλαμε επίσης η κατεξουσιοδότηση και οι εκτελεστικές πράξεις ε, να χρησιμοποιούνται λιγότερο στο privacy by design ή by default, που είναι ένα σημαντικό στοιχείο στην πρόταση του κανονισμού. Όπως επίσης και η ανωνυμοποίηση, ανονιμοποίηση των στοιχείων. Πολύ σημαντικό στοιχείο στο πλαίσιο των κοινωνικών δικτύων των δικτύων, κοινωνικής ε, δικτύωσης. Θα πρέπει να κάνουμε βέβαια περισσότερη δουλειά πάνω στους ορισμούς. Ένα άλλο σημαντικό κομμάτι της συζήτησής μας θα πρέπει να αφορά τη δικαιοδοσία και την ε, εφαρμοστέα νομοθεσία. Θα ήθελα εδώ να κάνω έναν παραλληλισμό μεταξύ του ρυθμιστικού, κανονιστικού πλαισίου και άλλων ρυθμιστικών ή κανονιστικών πλαισίων που εφαρμόζονται σε άλλες χώρες. Στις ΗΠΑ έχουμε το Patriot, Patriot Act, ένα νόμο που κάνει λόγο για την επεξεργασία των δεδομένων, επιχειρήσεως, οι έδρα των οποίων είναι στις ΙΠΑ. Ακόμη και αν έχουν γραφεία στην Ευρωπαϊκή Ένωση, για παράδειγμα. Υπάρχουν επίσης συμφωνίες μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και τρίτων χωρών σε σχέση με την διαβίβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, το PNR για παράδειγμα, η συμφωνία SWIFT. Οι συμφωνίες αυτές όμως ότι θα πρέπει να λαμβάνονται καλύτερα υπόψη στον κανονισμό. Μια άλλη σημαντική πτυχή αφορά τον ορισμό της σύμφωνης γνώμης, της συγκατάθεσης, θα πρέπει να είναι ρητή. Το consent. Δεν ε, ζητούμε βέβαια κάποια συγκεκριμένη μορφή για την χωρίς συγκατάθεση, για να μην προσθέσουν υπερβολική γραφειοκρατία στην όλη διαδικασία, αλλά θα πρέπει να είναι τόσο αναφερόμενη αυτή η έννοια και η συγκατάθεση ίδια. Μια άλλη σημαντική πτυχή είναι το δικαίωμα, αν θέλετε, στη λύθη ή στη θύμηση. Το να έχει κάποιο δικαίωμα να τον θυμούνται ή να τον ξεχάσουν. Όπως είναι αυτά τα, αυτές οι ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης. Είναι ένα παράδειγμα. Συμφωνώ με τον εισηγητή Κέλ για το ότι είναι ανάγκη να γίνει σαφής διαφορά, σαφής διάκριση καλύτερα μεταξύ του ελεγκτή και του επεξεργαστή των δεδομένων. Στην προηγούμενη οδηγία, στην παλιά οδηγία, ήταν σαφής η διάκριση αυτή. Στο νέο όμω κανονισμό είναι κάπως αμβλημένες οι διαφορές και πρέπει να το λάβουμε υπόψη μας αυτό. Πρέπει να πάρουμε τη σωστή απόφαση γιατί θα πρέπει να ορίζονται τα στοιχεία οι ξεκάθαρα και οι διάφοροι φορείς θα πρέπει να γνωρίζουν ε, τα καθήκοντα και τις υποχρεώσεις τους. Ό,τι αφορά τώρα συμβάντα ασφαλείας ε, και την κοινοποίηση τέτοιων συμβάντων, ε, τέτοιων περιστατικών, έχουμε λάβει διάφορες απόψεις από τον κλάδο που θεωρεί ότι είναι πολύ μικρή η προθεσμία του 24 ου για να ενημερωθούν οι χρήστες. Νομίζουν ότι θα είναι καλύτερο Ε, χρήστες φυσικά. Τα θύματα θα τα χαρακτηρίζαν να ειδοποιούνται, να ενημερώνονται, αλλά σημαντικό είναι και η αρχή να ενημερώνεται. το εντός ε, του 24ωρου δεν σημαίνει θα πρέπει να λυθεί και το πρόβλημα ή να βρεθεί το αίτιο. Για την κοινοποίηση μιλάμε, ότι ενημερώνεται και η αρχή και ο ενδιαφερόμενος για το γεγονός ότι υπήρξε διαρροή, κάποιο προσωπικού στοιχείου, προσωπικού δεδομένου. Αυτό είναι σημαντικό, γιατί το αν λόγω άτομο πρέπει να μπορεί να πάρει μέτρα προστασία. Θα σταματήσω εδώ και περιμένω τα σχόλια των συναδέλφων και τις απόψεις. Είμαι όμως βέβαιη ότι μέχρι στιγμής και θα συνεχίσουμε έτσι, έχουμε δουλέψει πολύ καλά. Φιώνα Χολ. Ευχαριστώ. κυρία Πρόεδρε, την κυρία Βαλιάν ε, από την Άλτε γιατί δεν μπορεί να είναι εδώ Ευχαριστούμε λοιπόν πρώτα απ' όλα τον εισηγητή για μια πάρα πολύ καλή γνωμοδότηση που αντιμετωπίζει τα περισσότερα από τα ζητήματα που απασχολούν τον κλάδο. Θεωρούμε πως ο εισηγητής βελτίωσε την πρόταση της ε, Κομισιόν με το να αντιμετωπίζει κάποια από τα ζητήματα πολύ λογικά και νομίζω πως μπορούμε να συνεργαστούμε πάρα πολύ καλά. Καλωσορίζουμε επίσης ε, την εστίαση στην αναλογικότητα καθώς έτσι θα επιτευχθεί η σωστή προστασία και από υπερβολικές, υπερβολικά γραφειοκρατικές διαδικασίες. Αυτό αφορά βεβαίως και τις διοικητικές κυρώσεις και τις παραβιάσεις και τις περιπτώσεις παραβιάσεων προσωπικών δεδομένων και ενισχύουν αυτή την πρόταση. Θεωρούμε πως ε, πρέπει να ξεκαθαρίσουμε τους ορισμούς για να μπουν τα πράγματα σε ένα σωστό πλαίσιο. Οι ορισμοί της συγκατάθεσης της κύριας έδρας και των ειδικών κατηγοριών ε, προσωπικών δεδομένων έχουν βελτιωθεί αρκετά. Επίσης θεωρούμε όσο ο σωστά αντιμετωπίζει τις πιθανές συνέπειες του κανονισμού όσον αφορά τους κλάδους της υγείας ε, και των χρηματοοικονομικών και θα πρέπει να μην δημιουργήσουμε περισσότερο διοικητικό βάρος χωρίς κάποιο συγκεκριμένο όφελος για τον καταναλωτή. Ξέρουμε πως ε, ήταν εδώ πέρα έντονες οι συζητήσεις όσον αφορά τον αριθμό και την έκταση των πράξεων κατά εξουσιοδότηση που προτείνει η Κομισιόν. Γι' αυτό καλωσορίζουμε τη ρεαλιστική προσέγγιση του κυρίου Κέλλη για την διαγραφή των περισσότερων από αυτών. Επίση, θεωρούμε πω θα μπορούσαμε να έχουμε πετύχει το κείμενο από την αρχή και να μην το αλλάζουν μετά η Κομισιόν. Και οι τεχνικέ προδιαγραφέ είναι ζήτημα βεβαίω που αφορά τον κλάδο και όχι την Κομισιόν. Στι τροπολογίε μα ελπίζουμε να δούμε κάποια από τα υπόλοιπα ζητήματα και προτείνουμε περαιτέρω βελτιώσεις οι οποίες θα συμπληρώνουν την γραμμή του εισηγητή. Θα εστιάσουμε στους ορισμούς ε, και στην διάκριση μεταξύ των ευθυνών των ελεγκτών και αυτών οι οποίοι επεξεργάζονται τα δεδομένα για να μην υπάρχει αλληλεπικάλυψη και όλοι να ξέρουν τι απαιτείται από αυτούς. Επίσης, σκοπεύουμε να δούμε το τι γίνεται με την φορητότητα των δεδομένων και τα προφίλ. Θα μπορούσαμε επίσης να έχουμε και άλλους ε, συγκεκριμένους, ε, συγκεκριμένες ανησυχίες. Θα δούμε λοιπόν τις ανησυχίες αυτές χωρίς να επιβαρύνουμε ιδιαίτερα τις ευρωπαϊκές εταιρείες και ειδικά τις μικρομισές επιχειρήσεις σε καιρούς κρίσης. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε. Αντεζότερ όδησα από τους Πράσινους. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε με έχει λίγο προβληματίσει αυτή η γνωμοδότηση γιατί δημιουργεί εξαιρέσει ε, για την προστασία των προσωπικών δεδομένων που θα είναι επιζήμια για την προστασία των δικαιωμάτων των φυσικών και νομικών προσώπων. Και επίση ό,τι αφορά τη μεθοδολογία έχει κάποιε προτάσει που δεν βρίσκουν απόλυτα σύμφωνοι. Αποδυναμώνεται έτσι η πρόταση και τελικά οι ιδιωτικά ε, φορεί ε, δεν έχουν τα απαραίτητα εργαλεία Δηλαδή δεν μπορούν να εξασφαλίσουν ε, ότι πράγματι υπάρχει προστασία. Και αυτό έρχεται σε αντίθεση με προηγούμενε τοποθετήσει του Κοινοβουλίου. Έχουμε πει δηλαδή εμεί συγκεκριμένα ότι δεν θέλουμε να αποδυναμωθεί η προστασία των δεδομένων. Πριν από ένα χρόνο είχαμε πει ξεκάθαρα ότι θέλουμε η προστασία των δεδομένων τουλάχιστον να είναι όσο ε, ισχυρή ήταν στην οδηγία του 1995. Φασίζουμε λοιπόν τώρα για το μέλλον της Ευρώπης και τις αξίες της. Ας το κάνουμε χωρίς να απεμπολίσουμε την ηθική ευθύνη μας προς τις εταιρείες, γιατί στην Ευρώπη είμαστε όλοι στο 2012. Έχω κάποιες άλλες ε, ενστάσεις. Για την τροπολογία 6 παραδοσιακά του κ. Κέλ που προτείνει να περιληφθεί το συμφέρον των τρίτων μερών. Αυτό έρχεται σε αντίθεση με κάποια δικαιώματα δεν μπορούν να δώσουν δηλαδή τη συγκατάθεσή τους αυτοί οι φορείς. Είναι ένα δικαίωμα που δεν έπρεπε να το είχαν. Καλύτερο θα ήταν αυτό το legitimate interest, το θεμητό συμφέρον ε, που είναι ο αντικείμενο αυτής της τροπολογίας, να το απαλείψουμε. Ελπίζω να με στηρίξετε. Τροπολογία 38. Προτείνω ο κύριος Κέλλη να μην μπορεί να αποσυρθεί από συμβάσει που έχει συνάψει ο με του ελεγκτέ. Η ελευθερία όμως για την ε, σύναψη ή τη λύση κάποια σύμβασης ε, νομίζω ότι πρέπει να διατηρηθεί. Άρα δεν μπορούμε να ειστερίξουμε. Τώρα για συστήματα ανθεκτικά και και από την πλευρά των εγκρίσεων γίνονται κάποιες προτάσεις από την τροπολογία 12 του κυρίου Κέλλη. Δεν είναι σωστή γιατί οι εμπειρογνώμονες από το τομέα της ασφάλειας μου έχουν πει ότι η προηγούμενη εμπειρία από τη ΣΥΠΑ με τις εν λόγω εξαιρέσεις δεν ήταν ικανοποιητική. Ο ορισμός της ανωνυμοποίησης επίσης θα πρέπει να βελτιωθεί. Γιατί θα μπορούσε να αφήσει κάποια παραθυράκια. Και αυτό πρέπει να το αποφύγουμε, γιατί θέλουμε να υπάρχει η μέγιστη ανωνυμοποίηση για αυτόν τον κανονισμό. Επίσης ένα προβληματικό τόσε πολλές εγκρίσεις και τόσε ε, πολλές ε, εξαιρέσει καταργούνται από τον κύριο Κέλλη. Και ξέρουμε και από το παρελθόν κάποιε εταιρείε ότι αποδυνάμωσαν τα επίπεδα προστασία ουσιαστικά. Άρα, εμεί θα πρέπει να περιλάβουμε αυτά τα έγγραφα και αυτέ τι εγκρίσει και όχι να τι απαλείψουμε. Επίση, θα ήθελα στην γνωμοδότηση να περιληφθούν και κάποια στοιχεία. Συμφωνώ για τη φορητότητα των δεδομένων. Πρέπει να διατηρηθεί. Αλλά την έχει αποδυναμώσει ο κ. Κέλλη. Και έξω και ενστάσει και από κάποιου φορεί του κλάδου. Δεν έχω πιστεί ακόμη λοιπόν ότι ισχυρισμοί σωστοί, τα φορητά δεδομένα είναι προσωρινά, παραμένουν προσωρινά και μετά την επεξεργασία τους και δεν σημαίνει ότι η επεξεργασία των δεδομένων από μόνη τη είναι φορητή, άρα δεν μπορεί να επηρεάσει τα επιχειρησιακά μοντέλα των επιχειρήσεων. Αυτό που γίνεται, αν αποδυναμωθεί η σχετική απέτηση για τη φορητότητα, είναι ότι δεν υπάρχει πλέον αυτονομία και έλεγχος αυτών των πληροφοριών. Άρα είναι το αντίστοιχο από αυτό που θέλουμε. Συμφωνώ επίση ότι είναι ε, ανάγκη να δουλέψουμε ακόμη περισσότερο την έννοια του δικαιώματο του να ξεχαστούμε. Όχι να συγχωρηθεί αυτό που θέλει να μην διατηρούνται τα στοιχεία του, δεν είναι το ίδιο. Δεν δηλαδή, θα πρέπει να δούμε ποιοι είναι αυτοί που έχουν μια συμβατική σχέση και για το significant Balance ε, θα πρέπει και αυτοί που ετούνται εργασία να ε, συμπεριληφθούν. Υπάρχουν πολλές ανησυχίες για, το, για τη σχέση αυτή και την ανισορροπία μεταξύ εργοδοτών και επίδοξων ε, απασχολουμένων. Πρέπει να το δούμε. Και καταπολέμηση του ντόπινγκ. Χαίρομαι που συμπεριελήφθη. Είναι σημαντικός και ο αθλητισμός και το ντόπινγκ. Η αρχική ε, πρόταση είχε αυτό το κενό και χαίρομαι πάρα πολύ που το διαβλέψατε. Αυτό με βρίσκει πολύ ικανοποιημένη, όχι βέβαια άλλα, άλλα σκέλη της πρότασής σας. Ευχαριστώ. Παρακαλώ δύο λεπτά όσοι λαμβάνουν το λόγο. Μας δυσκολεύει πολύ ο χρόνος. Πρέπει να ολοκληρώσουμε το πρόγραμμα. Βίνταλ Κουάντρας. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Η τελευταία σχετική νομοθεσία ευθύστηκε πριν από 17 χρόνια, οπότε έχει φτάσει η ώρα για μια επικαιροποίηση. Η πρόταση της Κομισιόν ε, σωστά τονίζει την ανάγκη για ένα πιο ξεκάθαρο συνεκτικό πλαίσιο το οποίο θα προωθεί την εμπιστοσύνη και δεν εμποδίζει την ψηφιακή οικονομία από την πλήρη ανάπτυξή της. Βεβαίως, αυτό πρέπει να αντισταθμιστεί από την ανάγκη προστασίας ε, των προσωπικών δεδομένων, την διασφάλιση της ιδιωτικότητας, της διαφάνειας και του σεβασμού των θεμελιωδών δικαιωμάτων. Εγώ συγχαίρω τον καλό μου φίλο, τον κύριο Κέλλη, για την έκθεσή του και συμφωνώ με τον στόχο του για να μειωθεί το διοικητικό βάρος για τις επιχειρήσεις. Έχουμε πολλές πρωτοβουλίες υποδιαμόρφωση για να τονίσουμε την ανάπτυξη και την απασχόληση ως προτεραιότητες ε, της ε, ευρωπαϊκής ε, βιομηχανίας. Και βεβαίως για να είμαστε συνεπείς με αυτή την πολιτική πρέπει να μην έχουμε γραφειοκρατικές διαδικασίες όπως οι διαδικασίες συνένεσης και της διατήρησης των αρχείων. Η συνένεση κάποιες φορές είναι ουσιαστική, αλλά κάποιες φορές δεν χρειάζεται. Όπως όταν ένας χρήστης έχει ζητήσει μία υπηρεσία η οποία απαιτεί προσωπικά δεδομένα. Αναφέρεται η ευρεία συνένεση και, και αυτή θα βοηθήσει να μειωθεί το βάρος. Επίσης, καλή ιδέα είναι να αναλύουμε τις εταιρείε οι οποίες έχουν ε, ενσωματώσει την λογοδοσία προστασίας προσωπικών δεδομένων και να μην τις τιμωρήσουμε με περαιτέρω διαδικασίες. Επίσης καλωσορίζω την ιδέα πως ευαίσθητα δεδομένα θα πρέπει βεβαίω σε περίπτωση παραβιάζονται να ε, σημαίνουν την επιβολή προστήμου. τίμου. Επίσης καλωσορίζω τον όρο ανωνυμοποιημένα δεδομένα και θεωρώ πως μέσω απλών τεχνικών βημάτων όπως τα ψευδόνυμα οι εταιρείε οι οποίες ε, βασίζονται σε αυτά όπως παραδείγματος χάρη έρευνα υγείας κτλ μπορούν να κάνουν τη δουλειά τους. Αυτά τα δεδομένα δίνουν δύναμη συχνά στον καταναλωτή, όπως παραδείγματο χάρη στην ενεργειακή αποτελεσματικότητα, ενώ τα στατιστικά στοιχεία μπορούν να δώσουν συγκριτικά στοιχεία για το πώς μπορούν να γίνουν αποτελεσματικότερα τα σπίτια των πελατών και πώς μπορούν να γίνουν σχετικές αλλαγές. Έχοντας αυτά κατά νου, θεωρώ πως θα είναι εποφελές να αναφέρουμε και τις εταιρείε αερίου και ηλεκτρισμού και τις εταιρείε δικτύου ενέργειας ως νόμους χρήστες και ελεγκτές προσωπικών δεδομένων που μπορούν να κάνουν χρήση του. Ευχαριστώ. Πιλάρ Καστίγιο. Πιλάρ Καστίγιο. Πρόεδρε, ευχαριστώ και γρήγορα γρήγορα. Εντάξει. Αυτή η μέση τη Επίτροπή, μάλλον για την οδηγία για Μα τα υπόλοιπα είναι κάτι το θετικό. Θα πρέπει να το βάζουμε σε ένα πλαίσιο ψηφιακό και χρειαζόταν ακριβώς ε, συγχαρτήρια στο Σον Κέλλη, το συνάδελφο, γιατί βοήθησε σε αρκετά σημεία και συζητιούνται, αλλά νομίζω ότι είναι θετικά, είναι ενδιαφέροντα αυτά τα στοιχεία μάλλον. Γι' αυτό ακριβώς σημαντικό θεωρώνε αυτά που λέει για ανώνυμα στοιχεία, τον ορισμό αυτών, τα ψευδόνυμα για διάφορες παραβάσεις των κανόνων ασφάλειας ή ακριβώς ε, επειδή πρόκειται για διαπιστευμένες ε, ενέργειες ε, την υπερβολική χρήση αυτών και εδώ θα πρέπει να δούμε τη διάκριση ανάμεσα σε ευθύνες ε, τι κάνει ο ένας και τι δηλαδή ο δηλαδή εκείνος που με διαδικασία και ο ελεκτής θα πρέπει να διατηρηθεί αυτή η απόφαση σημερινή οδηγία γιατί αυτή η πρόταση στα 26, 28 άρθρα και 29 επίσης ε, δημιουργούν σύγχυση για το ρόλο που παίζουν ε, αυτοί οι δύο ασχοληθεί με τη διαδικασία και αυτός που ελέγχει. Ο ελεκτής ε, λέει τι γίνεται με την όλη διαδικασία, ενώ εκείνος που ασχολείται με τη διαδικασία δεν έχει πρόσβαση σε αναγνωρίσιμα στοιχεία και ακόμη κάτι, νέες υποχρεώσεις σε αυτό που ακολουθεί η διαδικασία, όπως πάνω χάρη να κάνει διάφορες εκτιμήσεις, ε, ε, το τι, πώς τα πράγματα για προσωπικά στοιχεία, αλλά δεν μπορεί να προχωρήσει γιατί δεν γνωρίζει ακριβώς πώς έχουν αυτά τα προσωπικά στοιχεία, έχουν προσωπικό χαρακτήρα, έτσι. Και τρίτο κάτι, αυτός που έρχεται με τη δικασία, δηλαδή να, να πει και νέο ελεγκτής ώστε να μπορέσει να παρέμβει σε αυτά τα στοιχεία, αυτό συνδυάζεται άσχημα με τη δυναμική αυτής τις τεχνολογίες ε, της πληροφορίας επικοινωνίας στο ψηφιακό κόσμο, το σύστημα αυτό, ο κόσμο αυτό είναι ευαίσθητο, εύθραυστο, υπάρχει καινοτομία εκεί και αυτό. Και όμω αυτό χαρακτήρα θα πρέπει να διατηρείται παστησία κάθε στιγμή και σε σχετικά με αυτό που λέω, ίσω ε, θα μπορούσε να μπερδέψει ιδιαίτερα την όλη ανάπτυξη. Γι' αυτό ακριβώ να υπάρξει σημερινή διάκραση ανάμεσα σε αυτό που κάνει την ελεγχό και αυτό που ασχολείται τη διαδικασία, ο καθένα αρμοδιότητέ του, τα καθήκοντά του, εντάξει και τον ε, ολορισμό αυτών. Και τώρα το λόγο έχει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η Λάουρα Κορέντο, δόκτωρ Λάουρα Κοράντο, είναι παρούσα. Άκουσε, παρακολούθησε την σημαντική συζήτηση που έγινε, που διεξήχθη. Παρακαλώ λοιπόν θα μπορούσα να λάβει το λόγο. Ήθελα να ευχαριστήσω καταρχάς τον εισηγητή κύριο Κέλ για το σχέδιο εκθεσής του και βέβαια Πρέπει να πω ότι θα εξετάσουμε ε, το, την έκθεση ακόμη περισσότερο, ιδίω από το πρίσμα των σχολείων που έκανε ο ίδιο και οι υπόλοιποι βουλευτέ. Φυσικά και θα παρακολουθήσουμε τη συζήτηση που γίνεται και σε άλλε επιτροπέ. Την ΙΜΚΟ σήμερα, την ΛΥΠΕ και τι άλλε ενδεμένε επιτροπέ. Χαιρόμαστε που στηρίζει συνολικά του στόχου τη Κομισιόν το Κοινοβούλιο και τον ίδιο τον κανονισμό, τη μοναπιθετική θηρίδα, το One Stop Shop που εισάγουμε για να πλουστεύσουμε τα νομικά περιβάλλοντα για τις επιχειρήσεις. Είναι και ένας από τους βασικούς μας στόχους αυτός. Βέβαια, ένας άλλος στόχος είναι να ε, βελτιώσουμε το θεμελιώδης δικαίωμα της προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Έχουμε λοιπόν κατά νου και τους δύο αυτούς στόχους κατά την εξετάση αυτού του κανονισμού και ναι, πρέπει να βρούμε την ε, σωστή ισορροπία όπως υπόθηκε και από τον εισηγητή. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λοιπόν προτείνει αυτά που προτείνει για να ε, βρει τη χρυσή τομή Δηλαδή αφενός να βελτιώσουμε την, ε, τα δικαιώματα των προσωπικών δεδομένων και ταυτόχρονα να πλουστεύσουμε το νομικό περιβάλλον, να είναι πιο υπεύθυνοι οι υπόλογοι οι ελεγκτές, αλλά και να μειωθεί και το γραφειοκρατικό βάρος. Λάβω υπόψη μας τις ανησυχίες που εκφράστηκαν σήμερα. Ε, τις ε, ακούμε και από τα κράτη-μέλη και το Συμβούλιο για το διοικητικό αυτό βάρος και είμαστε ανοιχτοί από πλευράς Κομισιόν για να δούμε πώς μπορούμε να μειώσουμε ακόμη περισσότερο αυτά τα βάρη, τα διοικητικά. Αλλά χωρίς και να μειώσουμε ταυτόχρονα το επίπεδο της ατομικής προστασίας που είναι μια κόκκινη γραμμή για μας. Τουλάχιστον το ίδιο επίπεδο προστασίας να παραμείνει και βέβαια αυτό να προσαρμοστεί και στο επιγραμμικό περιβάλλον, στις προκλήσεις, στις δυνατότητες που διανοίγονται σήμερα για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων, κάτι που το 1995 δεν υπήρχε. Θα ήθελα να μιλήσω για την έννοια τη συνένεση, συγκατάθεση. Ε, επανήλθε και στην Επιτροπή ΙΜΚΟ σήμερα το πρωί. Είναι κάτι που ανησυχεί τα μάλα και τι επιχειρήσει, αυτή η ρητή συνένεση, συγκατάθεση. Η Επιτροπή θεωρεί ενίοτε ότι υπάρχουν ε, παρανοήσεις ε, ή τέλος πάντων δεν γίνεται αντιληπτή ακριβώς η έννοια αυτή, όπως την εννοούμε εμείς στην Κομισιόν. με την επέκταση έννοια για την επεξεργασία των δεδομένων. Θέλουμε να είναι ο βασικός στόχος, να είναι ο βασικός λόγος. Μάλλον θέλουμε να τη διευρύνουμε. Και βέβαια το θεμητό συμφέρον και τα λοιπά, όλα αυτά τα αίτια και οι λόγοι που υπάρχουν ήδη ε, θέλουμε να παραμείνουν όπως είναι σήμερα. Δεν έχουμε στόχο δηλαδή ούτε πρόθεση να δώσουμε προτεραιότητα στη ρητή συγκατάθεση για την επεξεργασία των στοιχείων. Όταν όμως χρησιμοποιείται η συγκατάθεση θα πρέπει να είναι καλή να έχει νόημα. Σήμερα αυτό δεν ισχύει. Η η αόριστη συγκατάθεση είναι μένει η οποία ερμηνεύεται και μεταφέρεται διαφορετικά στο εθνικό δίκαιο. Και κάποιες φορές όχι με το σωστό τρόπο. Θέλαμε λοιπόν να αυτή την έννοια διευκρινίσουμε και να πούμε ότι θα πρέπει να είναι πραγματική, όχι να είναι απαραίτητα γραπτή, γιατί αυτό δεν θα πει απαραίτητα ότι η ρητή είναι και γραπτή, Μιλάμε για οποιαδήποτε καταφατική δράση, ενεργητική ε, δράση εκ μέρους του ε, ατόμου. Τέλο πάντων να εκδηλώσει, να εκδηλωθεί με κάποιο τρόπο, εκδηλώσει αυτή την συγκατάθεση. Βέβαια υπάρχει και ισορροπία συμφερόντων ή και άλλοι λόγοι, συμβάσεις και τα λοιπά μπορούν να κινητοποιήσουν, να ενεργοποιήσουν τη διαδικασία της επεξεργασίας για να μην υπάρχει παρανόηση. Σας είπα τα σχετικά με την συγκατάθεση. Τώρα για τη φορητότητα και αυτό το σχετικό δικαίωμα είναι κάτι που το στηρίζει και ο συγητής και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι ανοιχτή στο να ε, διευκρινίσουμε το πεδίο αυτού του, αυτού του δικαιώματος. Το ίδιο και με αυτό δικαίωμα ε, στη λύθη που να ξεχαστείουν τα στοιχεία κάποια. Και εδώ πρέπει όμως να κάνουμε κάποιες περιττέρες διευκρινήσεις. Σταματήσω εδώ γιατί δεν έχουμε και πάρα πολύ χρόνο. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, επαναλαμβάνω, είναι ανοιχτή για να συνεχίσει τον επικοδομητικό διάλογο που είχε μέχρι τώρα και με το Κοινοβούλιο, με τον εισηγητή και με όλου του σκιώδει για αυτέ τι προτάσει. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ο συνάδελφος Κέλλη τώρα για να ολοκληρώσουμε τη συζήτηση αυτή την ενδιαφέρουσα. Ίσως και μερικά λεπτά μετά πέρα από αυτά που του στερήσαμε στην αρχή επειδή τον αγκάσαμε να επιταχύνει την παρουσίασή του. Εντάξει, εγώ θα είμαι σύντομος. Ήθελα απλά να ακούσω τι είχαν να πούν οι υπόλοιποι ομιλητές. Ενθαρρύνομαι συνολικά από τις παρεμβάσεις των συναδέλφων που δέχονται γενικά αυτά τα οποία λέμε και προφανώς ανισχούν βεβαίως. Εξάλλου πρόκειται μόνο για γνωμοδότηση. Γι' αυτό είναι οι γνωμοδοτήσεις για να τις συζητάμε. Νομίζω πως υπάρχει μια γενική ατμόσφαιρα ότι όλοι θέλουμε να επιτύχει αυτό το θέμα και για τους πολίτες και για τις επιχειρήσεις. Δεν ανέφερα τις πράξεις κατά εξουσιοδότηση Ναι, συνέστησα να ε, καταργηθεί, να καταργηθούν και τα είπε σωστά η Φιώνα Χολ. Είπε, εάν πετύχουμε το κείμενο δεν χρειάζονται πράξεις κατά εξουσιοδότηση. Άρα όσες περισσότερες τέτοιες πράξεις έχουμε δεν έχουμε κάνει καλά τη δουλειά μας. η Επίτροπος είπε πως υπάρχει ένα σημαντική πτυχή στο δικαίωμα να ξεχαστεί κανείς. Υπάρχουν αρχές, πρέπει να τις στηρίσουμε και να συμφωνήσουμε ίσως στο πεδίο εφαρμογή. Αυτό ελπίζουμε να κάνουμε. Ξέρω η Εμιλία ανησυχούσε και αυτό το καλωσορίζω. Όσον αφορά τις επιχειρήσεις. Το βασικό για εμένα είναι πως πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε να μειωθεί το διοικητικό βάρος. Δεν έχει νόημα να ε, φέρουμε περισσότερες ρυθμίσεις. Αυτή είναι η βασική πτυχή. Μία και μοναδική υπηρεσία επίσης είναι σημαντικό θέμα και τις υπόλοιπε πτυχές μπορούμε να τις δούμε ειδικά όσον αφορά τα ανώνυμα και ψευδόνυμα δεδομένα πολύ σημαντικά ζητήματα. Και νομίζω πρέπει να γίνει μια ευρεία συζήτηση από αυτόν για να μπορέσουν να υπάρξουν στις προτάσεις μας και ελπίζω να συμφωνήσουμε τελικά. Αναμένω λοιπόν τη συνεισφορά των συναδέλφων και την περαιτέρω συζήτηση. Δεν ξέρω, φαντάζομαι θα πείτε την προθεσμία για τροπολογίες. Ευχαριστώ. όπως προβλέπεται η οργάνωση του χρόνου. Δημόσια ακρόαση για που αποφάσισαν οι συντονιστές 17 Δεκεμβρίου από τις 4 μέχρι τις και 45 το απόγευμα βέβαια. Προθεσμία δε για την κατάθεση τροπολογιών 3η 18 Δεκεμβρίου μεσημέρι. Χωρίς μικρόφωνο η Ναι. Αυτά. Ανταλλαγή απόψεων τώρα. Για το stress test. Στην Ήτρε ακριβώς ψηφίσαμε 25 του μήνα μας πέρασε για μια προφορική ερώτηση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή να παρουσιάζαμε για τη δημοσίευση της ανακοίνωσης της Επιτροπής για το στρες, ε, για την έντονη πίεση λοιπόν. Προφορική ερώτηση αλλά και μία πρόταση ψηφίσματος της Επιτροπής Ήτρε. Για δώσουμε μια κατεύθυνση στη μελλοντική οδηγία για την ασφάλεια από τα πυρηνικά τον Ιανουάριο του 2013 κανονικά. Το σημερινό πρόταση ψηφίσματος είναι αποτέλεσμα συμφωνία ανάμεσα στι πολιτικές ομάδες. Όλα σχεδόν τα θέματα που παρουσιάστηκαν στο έγγραφο τη Επιτροπή τα καλύπτει. Θα σημεία που βρίσκουν αντίθετους θα συζητηθούν ε, κατά την παρουσία των ε, τροπολογιών. Όλες οι πολιτικές ομάδες 22 Νοεμβρίου είχαν τις μεταφράσεις στο κείμενο για να συντάξουν διάφορες τροπολογίες ενδεχόμενα και μετά μας πιέζει όμως ο χρόνος προθεσμία για τις τροπολογίες μέχρι αύριο το μεσημέρι. Τώρα το λόγο έχει, αυτό είναι και το πιο σωστό που θα πρέπει να κάνουμε, είναι τα διάφορα μέλη για να μπορέσουν να εκφράσουν τις απόψεις τους. Η συνάδελφος δικαστήριο πρώτη έχει το λόγο. Χωρίς πρόεδρο, χωρίς ε, μικρόφωνο. Uh, Ευχαριστώ. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να τονίσω την ε, συνεργατική προσέγγιση της ε, Προεδρίας ε, της Επιτροπής μας και νομίζω πως είναι πολύ ισορροπημένο το κείμενο της Προέδρου και αποτελεί μια πάρα πολύ καλή βάση. Πρέπει να τονίσουμε πως η αντίδραση στην Φουκουσίμα από την Κομισιόν και τις Εθνικές Ρυθμιστικές Αρχές για να λάβουμε μια πρωτοβουλία για αυτά τα stress ε, test έχει ήδη οδηγήσει σε κάποια ματά. Είναι συμπέρασμα ήδη πως δεν υπάρχει σοβαρή ανησυχία ασφαλείας ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Όμως, όμως τα τεστ αυτά κοπόσεως βρήκαν ε, αρκετά κενά όσον αφορά το επίπεδο ετοιμότητας σε εξωτερικά γεγονότα όπως οι πλημμύρες παραδείγματος χάρη. Ναι. Επίσης ε, αναφέρουν οι ρυθμιστικές αρχές πως όλα τα ενδιαφερόμενα κράτη-μέλη έχουν ξεκινήσει ή θα ξεκινήσουν εφαρμοστικές δράσεις για να κλείσουν τα κενά τα οποία βλέπουν. Ελπίζουμε λοιπόν να οδηγηθούμε σε κάποιες ελάχιστες προδιαγραφές ασφαλείας και ετοιμότητας σε επίπεδο Ευρωπαϊκή αλλά και από τις γειτονικές μας χώρες. Γιατί αλλιώς δεν ωφελούν τίποτα. Δεν πρέπει να επαναλάβουμε το περσινό λάθος, δηλαδή να γίνει μια συζήτηση υπέρ ή κατά της της πυρηνικής ενέργειας ή πώς θα γίνει τόσο ακριβή ώστε να μην είναι πλέον ανταγωνιστική. Θεωρώ πως πρέπει να επικεντρωθούμε στα τεστ αυτά και στα μαθήματα μπορούμε να αντλήσουμε για τη βελτίωση της πυρηνικής ε, ασφάλειας και ετοιμότητας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ιδεοδός θα βρούμε κάποια κοινά σημεία με βάση την έκθεση της κυρίας Σαρτόρη και δεν θα υπάρχουν ψηφοφορίε κλειδιά για καμία ομάδα. Έτσι θα μπορέσουμε να έχουμε ευρία πλειοψηφία και θα μπορέσουμε να στείλουμε ένα ισχυρό μήνυμα με τα συμπεράσματα μας στην Κομισιόν. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Χολ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ε, θα συμφωνούσα μαζί σας πως ήταν χρήσιμο αυτό το οποίο κάνατε, αλλά δεν ήταν αρκετά συνολικό θα έλεγα και έτσι στιβαρό. Είπε πως δεν υπήρχε ανάγκη να κλείσει κανένα εργοστάσιο, αλλά επίσης βρήκε πως ουσιαστικά όλα τα εργοστάσια πρέπει να βελτιωθούν και υπάρχουν διάφορα τεχνικά ζητήματα. Οπότε πρέπει κατηπηγόντες τα κρατη να δουν αυτές τις τάσεις και να εφαρμόσουν τις βέλτιστες πρακτικές που υφίστανται. Πρέπει να φροντίσουμε πως ε, οι αντιδραστήρες θα εφαρμόζουν τις πιο σύγχρονες πρακτικές που έχουμε. Και, όπως είπε η κυρία Ντελ Καστίγιο, κάτι τέτοιο δεν είναι φτηνό. Η Κομισιόν είπε πως το συνολικό κόστος των 132 αντιδραστήρων θα είναι γύρω στα 10 έως και 25 δισεκατομμύρια ευρώ τα επόμενα χρόνια. Αυτό το οποίο θα έλεγα εγώ είναι πως είναι σημαντικό η βιομηχανία, ο κλάδος να παραμείνει, να επιδείξει κάποια διαφάνεια για αυτό το κόστος. Δεν τίθεται ζήτημα επιδότησης και ελπίζω η Κομισιόν να χρησιμοποιήσει τις αρμοδιότητες της ε, στον τομέα του ανταγωνισμού και των κρατικών ενισχύσεων έτσι ώστε τα κράτη-μέλη να μην επιδοτούν τον κλάδο. Είναι ο μόνος κλάδος που υπάρχει πάνω από 60 χρόνια όπου το κόστος μονίμως ανεβαίνει αντί να πέφτει. Οπότε όσο και ζωτικές και είναι αυτές οι βελτιώσεις πρέπει ο κλάδος να επομιστεί το βάρος και να μην προσπαθήσει να κρύψει το ότι το κόστος αυτό είναι σημαντικό και απαραίτητο για τις διαδικασίες τους. Τέλος, κάτι το οποίο αφορά τη διαδικασία λήψης αποφάσεων. Η πυρηνική ενέργεια είναι μέρος ενεργειακής πολιτικής και της περιβαλλοντικής πολιτικής της Ένωσης και καθώς έχουμε αρμοδιότητες και σε άλλους τομείς και μπορούμε πραγματικά να έχουμε δικαιώματα συναπόφασης σε πάρα πολλά ε, ζητήματα, πρέπει να ξεκινήσει ένας επικοδομητικός διάλογος για τη μεταρρύθμιση της συνθήκης ΕΒΡΑΤΟΜ για να έχουμε και εδώ συναπόφαση. Είναι ανομαλία το ότι σε οτιδήποτε σχετίζεται με πυρηνική ενέργεια το Ευρωπαϊκό Κοινοβουλίο είναι εκτός. Ευχαριστώ, Μπαλτσιούτης. dėl Ευχαριστώ. Η ανακοίνωση της ε, Κομισιόν που αφορά την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων αυτών είναι κάτι το οποίο μας χαροποιεί και δείχνει πως η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει προβλήματα όσον αφορά την πυρηνική ασφάλεια. Τώρα, όσον αφορά τους μεγάλους κινδύνους και τα προβλήματα ασφαλείας, δεν μπορούμε να έχουμε διαφορετικές προδιαγραφές που θα ισχύουν σε κράτη-μέλη. Γιατί η πυρηνική ασφαλεία δεν αφορά μόνο το κράτος μέλος στο οποίο βρίσκεται ο αντιδραστήρας, γιατί ο αντίκτυπος ε, θα είναι αισθητό στο επίπεδο ολόκληρη Ευρώπης. Επίσης πρέπει να αντιληφθούμε το τι σημαίνει πυρηνική ασφάλεια. Ασφάλεια των υφισταμένων εγκαταστάσεων και αυτών οι οποίες ε, έχουν βγει εκτός. Να πω πως όταν βγαίνει κάτι εκτός, ε, βεβαίως μια τέτοια κατάσταση πρέπει να γίνουν πολύπλοκα έργα για τα εξαντλημένα καύσιμα που πρέπει να αποθηκεύονται για δεκαετίες. Οπότε πρέπει το ψηφισμά μας να περιλαμβάνει κάτι ε, σχετικό και για την ασφάλεια των εργοστασίων που έχουν κλείσει. Τώρα, το ζήτημα αυτό του κλεισίματος γίνεται πιο πολύπλοκο. Έχουμε προβλήματα που δεν τα είχαμε σκεφτεί και με τον κύριο βεβαίω θα γίνει ακόμη πιο δύσκολο και ε, πανηρώ. Γι' αυτό πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να παίξει έναν ηγετικό ρόλο και να παρουσιάσει προτάσεις σε σχέση με τις ε, αρχές ε, κλεισίματος ε, των υφιστάμενων τέτοιων εργοστασίων. Πρέπει να τα τονίσουμε όλα αυτά και ειδικά το ευρωπαϊκό επίπεδο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Μπρεζίνα. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι θα ήθελα να πω ότι αυτά τα τεστ αντοχής έγιναν ε, σε εθνικό επίπεδο, σε συνάρτηση με την αρχή της επικουρικότητας. Και οι ρυθμιστές ε, ήταν αυτοί που είχαν την απαιτούμενη εμπειρία για να φέρουν σε πέρα αυτούς τους ελέγχους. Με ιδιαίτερη χαρά διάβασα τα αποτελέσματα αυτών των ε, τεστ τα βλέπουμε και στους πίνακες που έχουν καταρτήσει οι εθνικοί ελεγκτές. Ωστόσο, υπήρξε ένα πρόβλημα. Δηλαδή, σε ορισμένε περιπτώσεις έγινε πολιτικό θέμα, πολιτικό ζήτημα. Για παράδειγμα, ο Επίτροπος Έτιγκερ, με έκπληξε άκουσα, να λέει ότι στην Τσεχία, στο Τεμελίν, θα πρέπει να γίνει επιθεώρηση Δεν νομίζω όμως ότι υπάρχει ε, ιδεολογικό τείχος που μας χωρίζει. Ουσιαστικά αυτό που μας χωρίζει είναι χώρες που χρησιμοποιούν την πυρηνική ενέργεια και χώρες που δεν χρησιμοποιούν πυρηνική ενέργεια. Και για να ε, δώσουμε τώρα πολιτικό χαρακτήρα σε αυτό, το θέμα δεν νομίζω ότι θα ήταν κάτι δίκαιο. Θα πρέπει όλες οι χώρες να αντιμετωπίζονται ισότιμα. Πρέπει να την εξασφαλίσουμε αυτήν την ισότιμη μεταχείριση. Γίνονται κάποιε διαφορετικέ ερμηνείε, ε, να αξιολογήσουν από κάποιου συμπρογνώμονε, οι προτάσει ε, των τροπολογιών που έχουν ως στόχο να δοθούν μεγαλύτερε εξουσίε στην Κομισιόν. Είναι κάτι με το οποίο δεν συμφωνώ. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Το Ζενόφσκι. Eh, Ευχαριστώ. Εγώ πραγματικά χαίρομαι πάρα πολύ που έγιναν αυτά τα τεστ αντοχής και που είδαμε ότι πραγματικά ε, τα πυρηνικά εργοστάσια μας ε, είναι σε πολύ καλή κατάσταση και δεν, εντάξει χρειάζεται κάποια να κλείσουν γιατί η ποιότητα των ε, ή πάντων αποτελέσματα δεν ήταν ε, τέτοια που να μας δίνουν σαφή ένδειξη για το τι πρέπει να γίνει με κάποιους, αλλά τέλος πάντων είναι πολύπλοκες εγκατεστάσεις, αυτές τις οποίες μιλάμε, αν αντίστοιχε ε, δοκιμές έγιναν σε άλλες εγκαταστάσεις, μη πυρηνικές, θα εκπληγόμαστε από τα, εκπλησόμαστε μάλλον από τα αποτελέσματα και θα βλέπουμε ότι ίσως να χρειάζεται να γίνουν αλλαγές από μια ώρα στην άλλη. Ελπίζω να βοηθήσει πάντως να ε, ηρεμήσει κάπως ε, η κατάσταση γιατί λεγόταν πριν ότι τα 5% των πυρικών σταθμών δεν πρόκειται να περάσουν τα τεστ και κάποιοι ανησυχούσαμε. Κάποιοι ανησυχούσαμε. Εγώ χαίρομαι πάρα πολύ με τα θετικά αποτελέσματα αυτών των ε, τεστ. Χαίρομαι επίσης ταυτόχρονα που βλέπω και ότι στα μεμονωμένα κράτη-μέλη αποδίδει και η πυρηνική εποπτεία. Είναι ανεξάρτητη και μπορεί να εκφράσει και κριτική. Φαίνεται να λειτουργεί σε αυτό το επίπεδο, όπως και στο εθνικό, μάλλον και στο ευρωπαϊκό και η συνεργασία. Οι διάφοροι οργανισμοί και φορείς έδειξαν ότι τελικά έχουμε ένα επαρκές σύστημα. Δεν βλέπω λοιπόν κανένα λόγο να αλλάξει αυτό το σύστημα των ελέγχων που έχουμε θεσπίσει σε εθνικό επίπεδο. Διότι φάνηκε ότι είναι ανεξάρτητο, ποιοτικό σύστημα, όπως ακριβώς το περιμέναμε. Αυτό που θα με ενσυχούσε, αντίθετα, θα ήταν αυτά τα καθήκοντα, οι αρμοδιότητες αυτές να μεταφερθούν σε ευρωπαϊκό επίπεδο και θα είχαμε πραγματικά πάρα πολλές αντιπαραθέσεις σε επαγγελματικό επίπεδο. Λοιπόν, εδώ έχουμε αυτό το stress test. Θα ήθελα να επιθυμίσω κάτι που συνέβη στην Ιαπωνία. Να τονίσω ότι πρόκειται... Είχαμε δύο φυσικές καταστροφές. Λοιπόν, το πρόβλημα δεν ήταν η πυρηνική τεχνολογία αλλά τα κενά όσον αφορά τον όλο σχεδιασμό, την όλη οργάνωση. Γι' αυτό ακριβώς ε, ο ρυθμιστής ο Ιάπωνας ε, και εκείνοι που διαχειριζόνταν το, τις εγκαταστάσεις δεν είχαν καμία έκθεση μετά για την ασφάλεια. Εδώ θα πρέπει να εκμεταλλευτούμε ακριβώς ευρωπαϊκές χώρες που έχουν ε, την καλύτερη αντιμετώπιση σε θέματα ασφάλειας για τα πυρηνικά τους εργοστάσια. Να λοιπόν, γιατί χρειάζονται αυτά τα stress test. Στο ψήφισμά μας προσπαθούμε να τονίσουμε ότι παντού αυτή η αντίληψη περί ασφάλειας στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι όσο γίνεται υψηλότερη, καλύτερη στο μάξιμουμ επίπεδο. Γι' αυτό λοιπόν χρειάζεται να δούμε εάν χρειάζεται, αν πετείται πραγματικά να συμπληρώσουμε την ομοθεσία και μετά να ακολουθήσουμε και τις πρώτες συστάσεις των εμπειρογνωμόνων, των ειδικών, να δούμε αν όλα αυτά είναι εφαρμόσιμα και σε ευρωπαϊκό επίπεδο θα πρέπει από κοινού να προσπαθήσουμε να εργαστούμε και στα διεθνή φόρουμ ώστε να πετύχουμε υψηλή προστασία πυρηνική και στις τρίτες χώρες γιατί η πυρηνική ενέργεια δεν γνωρίζει σύνορα φραγμούς. Και έτσι θα έχουμε άλλο ένα εργαλείο για να εγγυηθούμε την ασφάλεια. Σαν νομοθέτες εμείς τι θα πρέπει να κάνουμε. Να δημιουργήσουμε τις προϋποθέσεις ώστε να τρέφουν ε, οι πολίτες μας και εμπιστοσύνη απέναντι στη βιομηχανία που ε, διαθέτει πείρα. Είχε σχετικές εμπειρίες. Το know-how να μην το σπαταλήσουμε. Ευχαριστώ. Herzog. Uh, Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Αυτή τη στιγμή γίνεται μια συνάντηση Αρμενίας και Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και συζητάμε άρα και τα stress test ε, των παιχνικών εργοστασίων της Αρμενίας. Οπότε η πρωτοβουλία μας από ό,τι φαίνεται εξαπλώθηκε και εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν πρέπει λοιπόν να θυμόμαστε πως συμμετέχουν και άλλες χώρες εδώ πέρα. Να σας υπενθυμίσω και τη Φουκουσίμα. Και βεβαίως αγαπητοί συνάδελφοι πως δεν μπορέσαμε να υιοθετήσουμε ψήφισμα γιατί οι διαφορές μας ήταν πιο σημαντικές από ένα κοινό ψήφισμα. Τα Σας τα λέω αυτά γιατί ελπίζω πως ε, πρέπει να ελπίζω να υιοθετηθεί αυτή η έκθεση γιατί είναι πάρα πολύ σημαντική και για την ευρωπαϊκή κοινή γνώμη και άρα μπορεί να βελτιωθεί αν το Κοινοβούλιο υιοθετήσει μια γνωμοδότηση. Τώρα, γιατί δεν είναι καλό το κείμενο της Κομισιόν. Έλαβα πολλές επιστολές από τον κλάδο πως η Κομισιόν ε, δήλωσε πολλές φορές πως οι βουλευτές ζήτησαν προτεραιότητα ή μάλλον τον κατάλογο κατάταξης. Δεν ζητήσαμε εμείς κάτι τέτοιο οπωσδήποτε. Θυμάμαι που όλοι οι βουλευτές ανεξαρτήτως κόμματος είπαν ε, και ανεξαρτήτως άποψη για την ποινική ενέργεια είπαν πως δεν είναι σωστό κάτι τέτοιο είχαν προβλήματα με ένα τέτοιο κατάλογο. Πρέπει να το πω αυτό. Δεν ήταν η Επιτροπή μας αυτή η οποία ζήτησε κάτι τέτοιο. Πρέπει λοιπόν να είμαστε πολύ προσεκτικοί αλλά και σωστοί στην απόψή μας για ένα ζήτημα το οποίο πρέπει να παραμείνει υπό τη συνθήκη Ευρατόμ και την επικουρικότητα χωρίς να αλλάξουμε αυτή την συνθήκη ή τη νέα συνθήκη που θεωρούμε πως θα την αντικαταστήσει. Και επίσης μην ξεχνάμε πως και σε άλλες χώρες έχει αλλάξει η άποψη του κοινού για την πυρηνική ενέργεια. Οι χώρες οι οποίες ήταν υπέρ της πυρηνικής παρέμειναν και οι χώρες οι οποίες ήταν κατά παρέμειναν κατά. Θα ήθελα μόνο να πω πως τώρα εάν κλείσει ένα πυρηνικό εργοστάσιο στη Γερμανία τότε τα stress test για αυτά τα οποία κλείνουν χωρίς να βγαίνουν εκτός θα ε, είναι κάτι το οποίο θα δούμε στο μέλλον. Είναι μια νέα εμπειρία για όλους ε, του κλάδου και της πολιτικής. Πρέπει λοιπόν να είμαστε πολύ προσεκτικοί με αυτά τα οποία έχουν ε, κλείσει αλλά δεν έχουν βγει εκτός λειτουργίας. Ευχαριστώ. Γιατί είναι και αυτό ζήτημα ασφαλείας. Συνάδελφο Σόντι. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να σας συγχαρώ για την ε, Επιτροπή μας θα καταθέσετε ένα κείμενο για τη συζήτηση για να μπορέσει να αποφασίσει το Κοινοβούλιο για το δύσκολο αυτό θέμα. Το έχω πει και ενώπιον του Επιτρόπου. Η ανακοίνωση της Κομισιόν νομίζω ότι κατά πάσα πιθανότητα απέτυχε να αντικατοπτρίσει την ποιότητα των ελέγχων που διενεργούνται σε επίπεδο κρατών μελών. Όπως και άλλοι βουλευτές, νομίζω ότι δεν έχει καμία τεχνική και επιστημονική ικανότητα για να αντιμετωπίσει αυτό το πολύπλοκο θέμα η Κομισιόν. Με τους μηχανικούς που δεν νομίζω ότι μπορεί με τους ειδικού που έχει η Κομισιόν να ε, εκφέρει άποψη. Και άλλωστε γίνεται σε πολιτικό επίπεδο γίνεται ένα σημαντικό ε, διάλογος για την ενέργεια, την αλλαγή του ενεργειακού μείγματος κτλ. Εγώ νομίζω ότι δεν ξέρω πώς θα έχουμε συναπόφαση και μέσω ευρατών. Έχουμε τις ε, επιλογέ εκθέσεις Κίνα που ψηφίσαμε σήμερα. Εγώ νομίζω ότι θα πρέπει όλα αυτά τα θέματα να τα συνδέσουμε μεταξύ τους. Και ολοκληρώνω για το κόστος. Δεν πρέπει να μην υπάρχει πλέον διαφάνεια, θα πρέπει να υπάρχει διαφάνεια και να συμπεριλαμβάνεται όλο το κόστος. Δεν μπορεί να μας λέει ότι είναι η πιο φθηνή ενέργεια χωρίς να μας δίνει πλήρη ανάλυση του κόστους, περιλαμβάνει και του κόστους ασφαλείας, ε, αποξύλωσης, απορροπλισμού μονάδων, ε, επεξεργασίας, ε, χειρισμού των πάντων του, της μονάδας κτλ. Εμείς πάντως ό,τι αφορά τις δικές μας αρμοδιότητες ως παγκοδεσμικό όργανο έχουμε εκπληρώσει το ρόλο μας, αλλά σας συγχαίρω για την πρωτοβουλία αυτή γιατί έτσι είχαμε τη δυνατότητα να τα συζητήσουμε μεταξύ μας. Μπορεί να μην συμφωνούμε πάντα, αλλά ευτυχώ που καθένα μπορεί στο κράτο μέσα του κάθε χώρα να αποφασίζει για το ενεργειακό μείγμα. Και αρτικά. Ευχαριστώ. Κυρία Πρόεδρε, και εγώ θέλω να σας συγχάρω γιατί είναι πολύ σωροπημένο αυτό το κείμενο και είμαι πεπισμένη ότι όλες οι πολιτικές ομάδες δεν ε, θα αφήσουν ε, οι διαφορές τους ε, για το αν είναι υπέρ κατά της πυρηνικής ενέργειας να τις αποσπάσουν από το πολύ σημαντικό θέμα της ασφάλειας αυτών των πυρηνικό σταθμών. Το είπατε κι εσείς στο ψήφισμά σας. Είναι πολύ σημαντικό να υλοποιηθούν τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας και κυρίως οι συστάσεις που ακολούθησαν την ολοκλήρωση αυτών των τεστ αντοχής. Νομίζω επίσης ότι περιοδικά θα πρέπει να γίνεται αναθεώρηση ως κάθε 5 ή 10 χρόνια. Και εξίσου σημαντικό είναι αυτή η περιοδική αξιολόγηση να βασίζεται σε κοινά πρότυπα ασφαλείας. Οι διαδικασίες δηλαδή θα πρέπει να αρμονιστούν σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Βέβαια, πάντα πρέπει να εφαρμόσετε και η αρχή της επικουρικότητας. Και ένα τελευταίο στοιχείο. Πρέπει να είναι και επαρκές το εξειδικευμένο προσωπικό. Και να είναι και αρκετό στον αριθμό. Όχι απλά εξειδικευμένο θα πρέπει να μας απασχολήσει το θέμα της υπεργολαβίας. Η υπεργολαβία είναι παρκώς καταρτισμένη. Σε ορισμένε χώρε με έχω δει σε πυρηνικά εργοστάσια να εργάζονται πάρα πολλέ ώρε. Αυτό μπορεί να δημιουργήσει πρόβλημα στις συνθήκες ασφαλεία. Οι εργαζόμενοι σε ένα πυρηνικό εργοστάσιο δεν θα πρέπει να είναι από το ζυγό της λιτότητας ε, όπως ε, προκύπτει λόγω της οικονομικής κρίσης. Το προσωπικό ασφαλής πρέπει να προστατεύεται και γενικώ το προσωπικό των ε, πυρηνικών σταθμών από αυτή τη λιτότητα. Ευχαριστώ. Ο Σνάσου πρώτη τώρα. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Να τονίσω όπως και πριν ότι όλη τη διάρκεια ζωής ενός αντιδραστήρα θα πρέπει να καλύπτει ασφάλεια. Και θα πρέπει λοιπόν να λαμβάνουμε υπόψη μας και τα διάφορα στοιχεία για την ασφάλεια και το κόστος για τις επόμενες ενέργειες. Δηλαδή την διάλυση αυτού στο τέλος και πού πάνε τα απόβλητα τα πυρηνικά. Από το GRC έχει γίνει μια εκτίμηση το commercial είναι αυτό. Θα είναι κάτι το επίκαιρο και τα επόμενα χρόνια αυτός ο παροπλισμός και θα στοιχίζει περίπου 50 δισεκατομμύρια ευρώ. Θα πρέπει να το λάβουμε υπόψη μας. Και κάτι ακόμα. Εδώ λοιπόν θα πρέπει να δούμε τα διάφορα συστήματα ακριβώ που μας απασχολούν όσον αφορά το απόβλητα και επίση ο διοικό χαρακτήρα της πυρηνική ενέργειας οι στρατιωτικέ εφαρμογές αντί ακριβώ για να μειώσουν το κόστος όθησαν στην ε, υιοθέτηση της πυρηνικής ενέργειας και γνωρίζουμε το, τι επέφερε αυτό σαν αποτέλεσμα. Βίντελ Κουάντρας τώρα. Ναι. Καλωσορίζουμε αυτό το ψήφισμα. Ήταν αρκετά ουδέτερο για να το ο καλύτερος τρόπος ποιος είναι να είμαστε ουδέτεροι και αυστηροί και να αρκεστούμε ακριβώς στα γεγονότα και όχι ιδεολογικές ξεπερασμένες συζητήσεις πια. Τα γεγονότα ποια είναι. Η Ευρωπαϊκή Ένωση και μετά από το ατύχημα της Φουκουσίμα εμείς υποχρεωτικά ελέγξαμε με τεστ ε, της πυρηνικές μας εγκαταστάσεις και δείξαμε ότι η πυρηνική ενέργεια σε μας έχει προτεραιότητα. Εδώ για τις ε, ρυθμιστές ε, και τις εθνικές ρυθμίσεις ε, το ρόλο που έπαιξαν ήταν πολύ σημαντικός και είδαν ότι υπάρχουν και τομείς που μπορούμε να βελτιώσουμε την κατάσταση και ακριβώς το αρμοδιογραφείο υπέβαλε προτάσεις και ένα σχέδιο που θα μπορούσε να υιοθετήσει κανείς. Σίγουρα υπάρχουν περιθώρια να βελτιώσει κανείς την κατάσταση και ακριβώς όπως την ανακοίνωση αυτή της Επιτροπής αναγνωρίζεται από τα τεστ, από τις δοκιμές προκύπτει ότι δεν υπάρχει κανένας λόγος τεχνικής φύσεως για να κλείσει ούτε μία πυρηνική μας εγκατάσταση. Και έγινε μια διάκριση ανάμεσα σε δύο έννοιες που σε ορισμένε γλώσσες Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν υπάρχει διαφορετική λέξη. Υπάρχει το safety και το security στα αγγλικά. Και τα πρώτα είναι το nuclear safety και υπήρξε σύσταση μιας ομάδας εργασίας για να ασχοληθούν με το security, το δεύτερο. Και εκεί έχουμε ας πούμε και αεροπορικά ατυχήματα σχετικά. Έτσι, έχουμε nuclear safety και nuclear security. Θα πρέπει αυτά να συμπεριληφθούν στο ψήφισμα. Επίσης υπάρχει διεθνής νομοθεσία που ισχύει όσον αφορά την πυρηνική ασφάλεια, που σέβεται, πρέπει να σέβεται άλλωστε η Ευρωπαϊκή Ένωση. Και αυτή θα πρέπει να αναφέρεται σίγουρα στο ψήφισμα. Εντάξει, μπορεί να βελτιωθεί αυτό το τομέα, θα το επιθυμούμε, θα το προσπαθούμε, αλλά προ το παρόν να διατηρηθεί ω έχει, δηλαδή μια διαδικασία του Κοινοβουλίου σχετικά με την πυρηνική ασφάλεια και όχι κάτι το διαφορετικό. Το πνεύμα του ψηφίσματος θα πρέπει να το διατηρήσουμε, θα πρέπει να συνεχίσουμε την εργασία μας και να πετύχουμε ένα από τους κύριους και μόνιμους στόχους από τη στιγμή που υπήρξε η δημιουργία της Euratom και να έχουμε το ανώτατο δυνατό επίπεδο ασφάλειας και σίγουρα αυτό το ψήφισμα θα συνεισφέρει θετικά προς την επίτευξη αυτού του στόχου. Ευχαριστώ. Τελειώσαμε τις παρεμβάσεις και τώρα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει το λόγο. Επί του σημείου αυτού. Ναι. Για το stress test. Για να δούμε. Μισό λεπτό, μισό λεπτό, μισό λεπτό. Τούρμες. Ε, sorry ε, Με συγχωρείτε που άργησα. Το κείμενο νομίζω είναι καλή βάση, αλλά πρέπει να γνωρίζουμε πως το ζήτημα αυτό τεστ αυτό δεν ασχολήθηκε με σημαντικά ζητήματα όπως πτώσεις αεροσκαφών που εξετάστηκαν μόνο σε τέσσερις χώρες από πολύ περισσότερες που έχουν πυρηνικά εργοστάσια. Και βέβαια κάτι τέτοιο έχει νόημα αν στο τέλος υπάρχει κάποια κατάταξη. Και τολμήσουμε να πούμε, ε, εντάξει τώρα αυτοί οι αντιδραστήρες πρέπει να κλείσουν. Ούτε αυτό υπάρχει. Όταν λοιπόν συζητάμε το ποια θα πρέπει να είναι η επόμενη αναθεώρηση της οδηγίας και ένα άλλο ζήτημα πρέπει να δούμε είναι το ζήτημα της ευθύνης. Θα γνωρίζετε πως μετά τη Φουκουσίμα ο Ιάπωνας φορολογούμενος έχει να πληρώσει ένα λογαριασμό που υπολογίζεται στα 96 δισεκατομμύρια ευρώ τα οποία η εταιρεία δεν μπορεί να, να πληρώσει γιατί χρεοκόπησε, οπότε τα πληρώνει ο φορολογούμενος. Οποιοδήποτε μεγάλο πυρηνικό ατύχημα στην Ευρώπη θα το υπομειστεί ο φορολογούμενος. Αυτό είναι η λανθασμένη βάση που έχουμε σήμερα. Οπότε έχουμε μια εσωτερική αγορά ηλεκτρισμού, χτίζει κανείς π.χ. φωτοβολταϊκά ας πούμε, ε, πρέπει να πληρώσει την ασφάλιση να δώσει λεφτά για να βγάλει τις εγκαταστάσεις και τα λοιπά, ή αν είναι ολικά ας πούμε, όλα πρέπει να πληρωθούν. Και δεν με προκαλεί διοξίδιο του άνθρακα. Ε, όταν έχουμε διοξίδια, ε, ε όταν έχουμε πυρηνικά εργοστάσια δεν πληρούνται για τον κίνδυνο ούτε για τον παροπλισμό ούτε για τα απόβλητα και η μεγαλύτερη στρέβλωση στην εσωτερική αγορά προέρχεται από το ότι έχουμε αυτή την τεχνολογία η οποία για ιστορικούς λόγους ποτέ δεν ε, επομίστηκε το κόστος και αυτό είναι κάτι που πρέπει να αντιμετωπίσουμε στην οδηγία αυτή αν θέλουμε να είναι μια οδηγία η οποία θα μας βοηθήσει να έχουμε ίσους όρους ανταγωνισμού. Ευχαριστώ λέει και Πρόεδρος. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πρώτα απ' όλα να πω πως καλωσορίζουμε το σχέδιο ψηφίσματος γιατί όπως πολλοί είπαν είναι ισορροπημένο καλύπτει τις ε, πτυχές που είχαμε στην ανακοίνωσή μας όπως η εφαρμογή των συστάσεων που προέκυψαν από αυτά τα τεστ, ετοιμότητα για καταστάσεις εκτάκτου ανάγκης, αναθεώρηση της οδηγίας, ασφάλεια και αστική ευθύνη, καθώς και προσπάθειες να βελτιωθεί η διεθνής νομοθεσία. Να ξεκινήσω λέγοντας πως τα τεστ αυτά ήταν εθελοντικά και άνευ προηγουμένου στην Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί για πρώτη φορά ακολουθούσαμε την ίδια μεθοδολογία για να έχουμε μια ενιαία αξιολόγηση του κινδύνου όλων των πυρηνικών εργοστασίων. Εργαστήκαμε με την ENSREC και νομίζω πως το τελικό αποτέλεσμα ε, είναι πλέον αποδεκτό ως το διεθνές μέτρο σύγκρισης όσον αφορά τέτοιες αξιολογήσεις. Γι' αυτό θέλω να τονίσω την ιδιαίτερα θετική συνεισφορά και από την πλευρά των ρυθμιστών που υπολόγισαν πως ε, η προσπάθεια αυτή αντιστοιχεί σε 500 ανθρωποέτη και έγινε σε 18 μήνες. Θεωρώ πως η πρώτη προσπάθεια θα πρέπει τώρα να εστιαστεί στην εφαρμογή των συστάσεων. Δεν θα πρέπει να μείνουμε μόνο σε κάτι το οποίο θα μείνει στα χαρτιά στις Βρυξέλλες. Οι συστάσεις πρέπει τώρα να μεταμορφωθούν σε πραγματικότητα, σε επενδύσεις μέχρι το τέλος του έτους. Ε, μας έχουν υποσχεθεί πως ε, θα έρθουν στην Κομισιόν τα εθνικά σχέδια δράσης για να δούμε πώς θα ολοκληρωθεί αυτό. Συμφωνήσαμε με τις ρυθμιστικές αρχές να υπάρχει αξιολόγηση από τους ομότιμους και μετά θα πρέπει να δούμε πώς ακριβώς οι συστάσεις αυτές θα υλοποιηθούν η Κομισιόν γνωρίζει το ότι η φάση αυτή της εφαρμογής είναι εθνική ευθύνη όμως θα τα παρακολουθούμε από κοντά και όπως είπαμε στην ανακοίνωσή μας θα θέλαμε να υποβάλουμε μία αναφορά μέχρι τον Ιούνιο του 2014 και αν ενδιαφέρει το Κοινοβούλιο θα μπορούσε να τονίσει αυτή την υποχρέωση της Κομισιόν να δίνει αναφορά. Όσον αφορά δε τις περιπτώσεις εκτάκτου ανάγκης, ε, τονίσαμε αυτό το ζήτημα μαζί με τις ΜΚΟ και τις ρυθμιστικές αρχές ως προτεραιότητα και έχουμε ξεκινήσει μια μελέτη γι' αυτό. Όσον αφορά δε την αστική ευθύνη, όπως αναφέρθηκε, ε, εξακολουθούμε να αξιολογούμε την κατάσταση πιθανών θυμάτων και όπως είπαμε να αποφύγουμε και τους τις πιθανές τρευλώσεις του ανταγωνισμού στην ε, αγορά την ενιαία του ηλεκτρισμού που ελπίζουμε ότι θα υπάρχει μέχρι το 2040. Χαιρόμαστε ιδιαίτερα, κυρία Πρόεδρε, για το ότι καταφέραμε να έχουμε έντονες επαφές με τις γειτονικές χώρες και δύο από αυτές γειτονικές χώρες, Ουκρανία και Ελβετία, συμμετείχαν πλήρως στις δοκιμές. Οι άλλες ε, αποδέχτηκαν τη μεθοδολογία παρά ότι εφάρμοσαν διαφορετικά χρονοδιαγράμματα. Η διατύπωση για το ψήφισμα ε, για τη Λευκορωσία και τη Ρωσία ε, ίσως θα μπορούσατε να την ξαναδείτε γιατί είναι κάπως έντονη. Η Λευκορωσία δεν έχει ακόμα πυρηνικά εργοστάσια. Συμμετείχαν όμως σε όλες τις ε, συναντήσεις με την Ρωσία. Η Ρωσική Ομοσπονδία έχει ξεκινήσει δικά της εθνικά τεστ, αλλά δεν υποστήριξαν τη διαδικασία. Δεν υπέβαλαν δηλαδή εκθέσεις στους ομολόγους τους, αλλά απευθείας στην Διεθνή Υπηρεσία Ατομικής Ενέργειας. Τέλος, ε, σας διαβεβαιώ πως καταβάλουμε κάθε προσπάθεια για να βελτιώσουμε την εφαρμογή και πιθανή αλλαγή της ε, Διεθνούς ε, Πυρηνικής ε, Σύμβασης. Θα είμαστε βεβαίω σε όλες τις ομάδες εργασίας και όπως ακούστηκε δεν γνωρίζουν σύνορα τα πυρηνικά ατυχήματα, άρα αυτό έχει σημασία όχι μόνο εντός της Ένωσης αλλά και σε παγκόσμιο επίπεδο. Έχει δηλαδή σημασία να καταλήξουμε στο υψηλότερο δυνατό επίπεδο προστασίας. Και σας διαβεβαιώ πως, όπως ήταν ήδη προτεραιότητα πριν από το ατύχημα της Φουκουσίμα, η Κομισιόν θα συνεχίσει να ε, έχει την ποινική ασφάλεια ως ύψιστη προτεραιότητα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πολύ καλά. Να που ολοκληρώσαμε τη συζήτησή μας. Σας υπενθύμισα από την αρχή ότι ήταν ενδιαφέρον, σημαντικό να ακούσουμε και μεμονωμένα καθένα που πήρε το λόγο εκτός από τις ομάδες. Σας το υπενθύμισα όμως στην αρχή ότι μας πιέζει ο χρόνος και η προθεσμία για τις τροπολογίες είναι μέχρι αύριο την, την Τετάρτη μάλλον το μεσημέρι. Και παρακαλώ, αν μπορείτε να καταβάλετε αυτή την επιπλέον προσπάθεια. Αύριο Πέμπτη λοιπόν. Τελειώσαμε. Ξεκινάμε με τη συνάντηση των συντονιστών.